Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Θα ήθελα να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε όλες και όλοι στην ε, συνεδρίαση. Πριν περάσω στο θέμα υπαριθμών 2 της σημερινής διατάξεως, να σας ενημερώσω ότι ως συνήθως η συνεδρίασή μας μεταδίδεται από το διαδίκτυο. Σεις αποφασίζετε πώς ομιλείτε, αν χαμογελάτε ή όχι. Γιατί οι ψηφοφόροι θα σας παρακολουθούν. Θέμα 2 της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης έχει διανεμηθεί το σχέδιό της από 13ης πρώτου. Δεν έχω λάβει αιτήσει τροποποιήσεων, άρα θεωρώ ότι εγκρίνεται. Θέμα 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση. Οι συντονιστές θα επανέλθουμε στις 2.30. Ένα θέμα θα αναβληθεί για παραπέρα συζήτηση με την νομική υπηρεσία για άλλη συνάντησή μας. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα κάνουμε και με γραπτή διαδικασία. Ανακαλύψουμε ότι αυτό είναι δυνατόν. Αν δεν έχετε λοιπόν ε, πρόβλημα σχετικά, αυτό θα κάνουμε και θα τα ξαναπούμε ως Επιτροπή στις 3 το απόγευμα. Δεύτερη ανακοίνωσή μου, αποφάσεις που λήφθηκαν όσον αφορά τον διορισμό εισηγητών. Το Λαϊκό Κόμμα διόρισε τον Έστεμπαν Κονσάλες Πόνς ως εισηγητή για τη γνωμοδότηση για την συμφωνία TTIP η υπεύθυνη επί της επιτροπή είναι η ΙΝΤΑ. Οι σοσιαλδημοκράτες τον κύριο Ατόντο για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπεύθυνη ΛΥΜΠΕ, η ομάδα ECR τον κύριο Ουζαντόφσκι ως εισηγητή για γνωμοδότηση για τις αιτήσεις εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και αναλογικότητα, όπου αρμοδία της Επιτροπή είναι η νομικών υποθέσεων. Υπαριθμόν 4. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως. Τώρα για λόγους που δεν γνωρίζω ακόμη, γνωρίζουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση με τα πρακτικά. Σήμερα λοιπόν εγκρίνουμε τα πρακτικά της 6ης Οκτωβρίου. Μας μένει ακόμα Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Πάντως είναι διαθέσιμα τα πρακτικά και θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν υπάρξει ένσταση, πριν από το τέλος της συνεδριάσεως. Θέμα 5. Η κυρία Γκουλάρ είναι παρούσα. Έχουμε τη γνωμοδότηση της Σιλβί Γκουλάρ για λογαριασμό της ΕΚΟΝ επί του θέματος επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και οι σκιώδεις ηγητές επίσης είναι παρόντες Σιλβή. Σας ευχαριστώ, Ντανούτα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για αρκετά σημαντικό εγχείρημα. Βέβαια, χρειάζονται και ταλέντα συγγραφής, διότι είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός λέξεων και επομένως είναι σύντομη γνωμοδότηση. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της προτάσεως που θα σας κάνω. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, ότι τα θέματα της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης είναι τόσο σημαντικά, ώστε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε θα είναι, πρέπει να επιφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και το στοιχείο του κράτους δικαίου. Γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να πιστούν και πάλι οι πολίτε ότι τα όσα πράττουμε εδώ ανταποκρίνονται τουλάχιστον στι δημοκρατικέ παραδόσεις. Υπάρχουν διάφορα θέματα όπως είπα, δημοκρατική νομιμότητα, διαθεσμική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ώστε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων. Είναι κάτι το οποίο ζητεί ξανά και ξανά η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έχουμε και μια παράγραφο που λέμε ότι η δέσμη των έξι μέτρων που προβλέπει τον οικονομικό διάλογο, μα τι είναι ο οικονομικός διάλογος, είναι η ιδέα ότι όταν πρόκειται για μέτρα ή αποφάσεις σημαντικά για μια χώρα μέλος μπορεί να προσκληθεί ο Υπουργό Οικονομικών της χώρας αυτής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ Ευρωπαϊκού και Οικονομικού επίπεδου και Εθνικού επίπεδου να μην είναι μοναχά ο λόγος που εκφράζουν οι Υπουργοί Οικονομικών μέσα στη χώρα τους χωρίς να ακούγεται και η ευρωπαϊκή πλευρά και χωρίς να επωφελούνται και από την υποστήριξη που θα βρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, όπως είπαμε, στα πλαίσια της δέσμης 6 μέτρων που είναι πλέον νομοθεσία και που πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να αξιολογηθεί. Τώρα μια άλλη παράγραφος για την διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την οικονομική διακυβέρνηση. Το ερώτημα εδώ είναι πώς βλέπουμε τις σχέσεις μας με τα εθνικά κοινοβούλια υπό την έννοια ότι ο καθένας είναι πεπισμένος εδώ, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβουλία, διότι είναι φορείς νομιμότητας που δεν μπορεί να λυθεί κανείς. Και κάθε συνάντηση του Ευρωκοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν σημαίνει ότι αρκεί για να ε, ενισχυθεί η λογοδοσία. Αυτό και πολλοί εδώ έχετε αγωνιστεί υπέρ αυτό τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται ανάληψη ευθύνης όχι απλές συμπαθητικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που σίγουρα αποδίδουν, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά. Και ότι επομένω είτε παραμένουμε σε ένα επιφανειακό επίπεδο, είτε προχωρούμε στη δημιουργία ενός μεικτού οργάνου. Αλλά τότε πώς θα λειτουργήσει το όργανο αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι βουλευτές, οι εθνικοί βουλευτές δεν έχουν την ίδια βαρύτητα διότι προέρχονται από χώρες που η συνεισφορά του στο σύστημα δεν είναι ίδια. Ούτε μπορούμε να δεχθούμε ότι ορισμένα κοινοβούλια είναι πιο ισχυρά από άλλα. Αν το δεχθούμε αυτό θα φτάσουμε σε δυσκολίες. Από τη δική μου πλευρά δεν θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεικτά όργανα αλλά με ξεκάθαρες ευθύνες. Οι βασικές αυτές γενικές αρχές που ε, ανακοινώνουμε εδώ είναι δύσκολο να μπουν σε ένα σύντομο κείμενο. Εξάλλου έχουμε μια αναφορά στην επικαιρότητα, διότι είδαμε στην τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στα πλαίσια του σχεδίου Juncker ότι η Επιτροπή λαμβάνει την οδό, λαμβάνει δηλαδή και υπόψη και τις επενδύσεις στην αξιολόγηση που κάνει των εθνικών προϋπολογισμών. Έχει κάνει λοιπόν ένα βήμα η Επιτροπή που επιτρέπει στις χώρες να αφαιρέσουν από, τον, ε, από τους λογαριασμούς τους τις επενδύσεις που κάνουν κατ' εφαρμογή του ε, σχεδίου Juncker και τις ευρωπαϊκές συγχρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω πρέπει να πάμε λίγο πιο μακριά και να δούμε ποιες είναι οι επενδύσεις που μεσοπρόθεσμα μεν αυξάνουν το εγχώριο προϊόν των χωρών, αλλά δεν θέλουμε να οθήσουμε τις χώρες σε κακή εφαρμογή των κανόνων, αλλά με απασχολεί πολύ η επιλογή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Επιτροπή και λέει ότι έχουμε κανόνες επενδύσεις επί του Εθνικού ΑΕΠ, αλλά σας επιτρέπουμε να αφαιρέσετε τα όσα πηγαίνουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο που δεν θα αυξήσουν το ε, εθνικό εισόδημα το εθνικό προϊόν. Πρέπει να δούμε τις χώρε μέλη οι οποίε θα ζητήσουν τότε τη δίκαιη επιστροφή από το σχέδιο ε, Juncker. Γιατί βάζουν λεφτά σε ένα κοινό καλάθι ενδεχομένω όμως και για εθνικού λόγους. Και φοβούμε ότι θα δούμε αυτό που είδαμε και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, όπου αυτή η ιδέα τη δίκαιη επιστροφής έχει μολύνει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και εν τέλει θα μειωθούν οι επενδύσεις κατά το σχέδιο Juncker. Γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχει πρώτα ανάγκη να γίνει μια δουλειά για να ξεκαθαριστούν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, να μην ανοίξουν παράθυρα για καταχρήσεις, αλλά να μειώσουμε τις επενδύσεις που θεωρούμε ότι θα αυξήσουν το προϊόν. Είναι ορισμένε ιδέες που χρειάζεται κάπως, μεγαλύτερη ε, ανάπτυξη. Ήδη από την συνθήκη της Μάστριχτ δεν επεμβαίνει το δικαστήριο. Όμως ξέρουμε όπως έχει ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι από τους πιο σημαντικούς φορείς της ολοκλήρωσης και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πηγή δικαίου είναι το γεγονός ότι υπάρχει και κοινή δικαιική τάξη. Άρα μέτρα που εισδύουν βεβαίως και στην πολιτική των χωρών μελών, αλλά υπάρχει και ένας ανώτατος διαιτητής που είναι το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ υπάρχουν δύο οδοί δυνατές αυτή που επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να έχει κυριαρχία επί του Ευρωπαϊκού Δικαίου και που είναι η διαδικασία προσφυγής λόγω παράληψης και η προσφυγή για κατάργηση αποφάσεων του Συμβουλίου ή συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την ώρα δεν έχουμε το υλικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Είμαι όμως πεπισμένοι ότι για χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, που δικαίως και βεβαίω αποτείω φόρο τιμής στα όσα έπραξαν οι Γερμανοί, που είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στον δικανικό έλεγχο και στο κράτος δικαίου, θα ήταν επικίνδυνο να συνεχίσουμε ωστόσο με ένα σύστημα που βλέπουμε καθαρά ότι επινοούνται κυρώσει και που αυτέ δεν εφαρμόζονται. Πάντω δεν είναι αμεσοπρόθεσμο το θέμα αυτό. Όμως άπτεται τις θέσεις των ε, οργάνων απόδοσης δικαιοσύνη μέσα σε ένα πλαίσιο όπου οι νόμοι από το 1950 και 1957 λένε ότι μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιθέτως. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ακούω βεβαίω τις απόψεις όλων των άλλων εισηγητών και σχεδόν εισηγητών για να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση και δημιουργική και τολμηρή της Επιτροπής Συνταγματικών υποθέσεων. Χαίρομαι που είναι παρουσία και η Περβάμ Μπερέ. να δούμε πώς η γνωμοδότηση θα μπορέσει να ενταχθεί στην ε, ίδια την έκθεση που κάνει η ίδια για την αρμόδια επιτουσίας επιτροπή. Ναι, θα περάσουμε τώρα στους ε, σκιώδεις Για το, για το Λαϊκό Κόμμα υπάρχει κανεί, Όχι, από του σοσιαλιστές. Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Σιλβί Γκουλάχ για αυτή τη δουλειά που έκανε έτσι ώστε να μας δοθεί ευκαιρία εδώ στην ΑΦΚΟ να καταλήξουν σε μια κοινή, τολμηρή και δημιουργική θέση σε σχέση με αυτό το ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης. Η δική μας συνεισφορά θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο ε, της συνολικής προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ασιών της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της έκθεσης της κυρίας Μπερές. Η δική μας συνεισφορά λοιπόν, κατά την άποψή μας, Και σύμφωνα με τα όσα είπε η Σιλβή, θα πρέπει να είναι να υπογραμμίσουμε τις πολιτικές διαστάσεις της οικονομικής διακυβέρνησης. Και εδώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την αξιολόγηση που κάνει η έκθεση σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική νομιμοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Δημοκρατική νομιμοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει ένα σοβαρό ρόλο ε, στην εξασφάλιση αυτής της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Στο σχέδιο γνωμοδότησης όμως υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν μερικές επιφυλάξεις. Πρώτον, σε ό,τι αφορά ακριβώς την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη δεύτερη παράγραφο προτείνεται να συναυθεί, μάλλον να ε, καταστεί δυνατή η κοινοβουλευτική επικύρωση των διαφόρων σταδίων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα έπρεπε να διευκρινίσουμε τι ακριβώς εννοούμε αυτή την επικύρωση, αυτή, αυτή η, η λέξη δεν έχει σαφές νόημα. διότι δεν είναι γνωστή στο πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρόκειται για τη διαδικασία συναπόφασης. Ποια είναι η φύση αυτής της παρέμβασης του Κοινοβουλίου. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε επικοδομητικοί στην παρέμβασή μας, αν θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν καλό να είμαστε πιο σαφείς σε ό,τι αφορά αυτή την παρέμβαση. Μετά. Δεύτερο μου σχόλιο, επιφύλαξη. Γίνεται αναφορά στην συνθήκη της Λισαβόνας και στις δυνατότητες που ανοίγει σε ό,τι αφορά το θέμα των επενδύσεων. Η Σιλβία ακόμα και προφορικά είπε ότι θα πρέπει να υπερβούμε το όριο που έθεσε η Κομισιόν. Νομίζω ότι το σχέδιο νομοδότησης της ΑΦΚΟ θα πρέπει να ε, επικαιροποιηθεί υπό το φως των πιο πρόσφατων εξελίξεων των παρεμβάσεων της Κομισιόν. Για παράδειγμα, στο θέμα των επενδύσεων, αντίθετα με τα όσα αναφέρει η Σιλβή, αυτό που προτείνει δεν ξεπερνάει αυτό που λέει πλέον η Κομισιόν. Αντίθετα, υπολείπεται αυτόν που προτείνει η Κομισιόν πλέον. <laughs> Εγώ, για την ακρίβεια, συμφωνώ περισσότερο με αυτά που μας είπε η Σιλβή προφορικά παρά με όσα γράφονται στο έγγραφο της ε, νομοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τις δυνατότητες που ανοίγει η συνθήκη της Λισαβόνας ε, και μάλιστα σε διάφορα επίπεδα. Ένα από τα διδάγματα από την ευρωπαϊκή ε, κρίση είναι ότι καταπίπτουν πολλά από τα δόγματα που είχαμε, τα οικονομικά δόγματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη ε, να αρχίσει να αγοράζει ε, κρατικά ομόλογα, κάτι που αρνείτο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Επίσης, πλησιάζουμε σε ευελιξία σε ό,τι αφορά την ερμηνεία ορισμένων όρων, δημοσιονομικών όρων και κανόνων που παλιότερα ε, ήταν ταμπού. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει και με τις επενδύσεις και θα ήταν λάθος η ΑΦΚΟ να ε, στείλει ένα μήνυμα ε, το οποίο θα υπολείπεται των προτάσεων της Κομισιόν σε τέτοια το θέμα των επενδύσεων. Γιατί η Σιλβή στην έκθεσή της κάνει μια διάκριση ανάμεσα στα τρέχουσες δαπάνες και στις παραγωγικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να παράγουν συγκεκριμένο ε, αποτέλεσμα. Η Κομισιόν λέει κάτι παραπάνω από αυτό. Λέει ότι οι επενδύσεις δεν θα προσμετρώνται στο έλλειμμα και υπό όρους που ξεπερνούν τους όρους που θέτει η Σιλβή στην έκθεσή της. Οπότε ας μην παραμείνουμε ε, πιο πίσω από τις προτάσεις Κομισιόν. Ε, το θέμα αυτό έχει σχέση με την συνθήκη και με την ισότητα των κρατών σε ό,τι αφορά τη συνθήκη. Η Κομισιόν προτείνει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο καθεστώς που θα εφαρμόζεται στα κράτη ε, του τα ονομαζόμενα προληπτικού μηχανισμού ε, και στα υπόλοιπα. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε μνημόνιο και άλλες όχι. Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται σε μηχανισμό ελέγχου του ελλείμματος και άλλες όχι. Όμως θα πρέπει κατά την άποψή μου όλες οι χώρες να τη χάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Ε, και αν κάνουμε κάποια διάκριση, θα πρέπει η διάκριση να είναι αναλογική με τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, το κατά πόσον μπορεί η πρώτη Κομισιόν να προσαρμοστεί στην αρχή της ισότητας. Τώρα, σε ό,τι φορά αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με τις επενδύσεις για κοινωτικά σχέδια. Η Κομισιόν κάνει μια διάκριση ανάμεσα στις χώρες που βρίσκονται στο προληπτικό, σε προληπτικό στάδιο και στις χώρες που βρίσκονται σε διορθωτικό στάδιο. Στην, ε, στις χώρες που βρίσκονται στην πλευρά, τη διορθωτική πλευρά του συμφώνου, μόνο οι επενδύσεις ε, μέσω του ταμείου, ε, Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου δεν προσμετρώνται στο έλλειμμα. Ε, για τι άλλε χώρε θα προσμετρώνται στο έλλειμμα. Αυτή η διάκριση που κάνει η Κομισιόν εξηγείται από την διαφορά στο ε, θέμα του υπερβολικού ελλείμματος. Υπάρχει λοιπόν μια ανισότητα στη μεταχείριση η οποία δεν βασίζεται στις, ε, σε πραγματικές διαφορές. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα η κυρία Γκουλάχ να το δει. Τελευταίο σχόλιο για την παράγραφο 6 του σχεδίου νομοδότησης της ΣΥΛΒΗ. Ε, λέγεται εκεί ότι η ΑΦΚΟ εκτιμά ότι μια αναθεώρηση των συνθήκων περιορισμένης εμβέλειας ε, θα επέτρεψε το δικαστήριο να επιβάλλει κυρώσει. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την παράγραφο. Ε, το να ε, παραχωρήσουμε στο, Ευρωπαϊκό, δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις για ε, ε για τις παραλήψεις, είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί αναθεώρηση περιορισμένης εμβέλειας. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα η Σιλβή να διαγράψει αυτή την έκτη παράγραφο. Ευχαριστώ. Thank you, very much. Ευχαριστώ, Πέδρο. Ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι. Ε, το θέμα είναι τρομερά ελκυστικό, αλλά δεν έχουμε και άπειρο χρόνο. Ο Μάρκος είναι εδώ. Ο Πασκάλ είναι εδώ. Α, είστε εδώ. Συγγνώμη. Μιλώ εκ μέρου του Πασκάλ Ντιγόν που δεν είναι εδώ να παρουσιάσει την έκθεσή του. Λυπάται που δεν είναι εδώ μαζί μα. Πέντε σύντομα σημεία στην παρέμβασή του. Πρώτον, ευχαριστούμε τη Σιλβί Γκουλάχ για την πολύ καλή συνεισφορά της. Δύο, είναι σημαντικό να υπάρξει δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση μέσω της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλουμε διακυβερνητικές συμφωνίες σε αυτό το θέμα. Όχι. Τρίτον, είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε ποιες επενδύσεις δεν θα πρέπει να προσμετρώνται ως ε, δημοσιονομικό έλλειμμα. Δεν μιλάω μόνο για τις ε, παραγωγικές επενδύσεις. Εξάλλου είναι μια πολύ αόριστη έννοια η παραγωγικότητα, αλλά και σε κάποιες επενδύσεις που αφορούν την αλληλεγγύη με σκοπό να παράγουν αποτελεσματική ευημερία και πρόοδο για τους πολλούς. Τέταρτον, για την παράγραφο 4 και την δια... κοινοβουλευτική διάσκεψη. Η εμβέλεια και η έννοια αυτής της διάσκεψης θα πρέπει να διευκρινιστεί, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα εθνικά κοινοβούλια παίζουν ένα πιο σημαντικό ρόλο και ένα πιο διαρθρωμένο ρόλο. Πέντε για την παράγραφο 6. Εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα και σοβαρότατη διαφωνία. Το να διαγραφεί η παράγραφος 10 του άρθρου 126 με αυτή την απαλληφή ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Είναι πολύ υψίστος πολιτικό θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί με πολιτικό τρόπο. Εξού και η πρωτοβουλία δεν μας φαίνεται θετική. Αναγκοινώνουμε ότι η πράσινη ομάδα μας θα προτείνει τροπολογίες στα εξής τρία σημεία. Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, επικρίσεις του Eurogroup και της ε, Ευρωσυνόδου για το ότι σφετερίζονται νέες αρμοδιότητες χωρίς καμία νομική βάση και την εισαγωγή, την, ε, της εισαγωγής της ε, Κομισιόν για τις δράσεις της ως μέλος της Τρόικα. Ευχαριστώ, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Um, opinion. Uh, Χαιρετίζω την γνωμοδότηση της Σιλβή. Συμφωνώ με πολλά από τα σημεία και με πολλά από τα σημεία των συναδέλφων που μίλησαν για τη σημασία της παραγράφου μιλάει για την δημοκρατική λογοδοσία, που είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό και εμείς να πούμε ότι η διακοινοβουλευτική διάσκεψη είναι μια διάσκεψη όχι μόνο για τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά για τη βελτίωση της διακοινοβουλευτικής συνεργασία, συνεργασίας. Η νομιμοποίηση αυτή, η δημοκρατική νομιμοποίηση, θα πρέπει να δοθεί στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσει. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Για τι δύο τελευταίε παραγράφου. Καλωσορίζω το, τις γενικές διατυπώσεις για την πιο ευνοϊκή μεταχείριση των επενδύσεων στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Αλλά αυτό θα πρέπει να τεθεί σε ένα πλαίσιο με την ανακοίνωση για την ευελιξία ίσως οι απόψεις μας εδώ δεν είναι οι ίδιες. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση αυτή είναι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και δεν βλέπω πού υπάρχει το πρόβλημα με το σχέδιο Juncker. Γιατί στη νέα ρήτρα επενδύσεων ε, η συγχρηματοδότηση που προβλέπει ο Juncker είναι μία από τις δυνατότητες. Έχουμε και όλοι και έχουμε και το Ταμείο για τις υποδομές ούτως ή άλλως. Μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη ρήτρα ε, που βρίσκονται στο διορθωτικό βραχίωνα, στο βαθμό που αυτή η ρήτρα επενδύσεων βασίζεται στο άρθρο 1 του 1466 που αφορά τις ε, διορθωτικές επενδύσεις και που έχει επεκταθεί και σε χώρες ε, για το διορθωτικό βραχίωνα. Επομένως, λογικά και νομικά, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τη ρήτρα επενδύσεων. Θα πρέπει να καλωσορίσουμε την ανακοίνωση για την ευελιξία και νομίζω θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και χώρες σε αυτή την ρήτρα επενδύσεων ε, που βρίσκονται στο διορθωτικό βραχίωνα. Ε, συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους για τις αμφιβολίες που έχουν για την παράγραφο 6 για δύο λόγους. Καταρχάς, το ενιαίο νόμισμα απαιτεί μια οικονομική πολιτική. Όχι μια απλή, ένα απλό αυτοματοποιημένο κανόνα που να προχωρήσει τη διακυβέρνηση. Η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να συνδέεται περισσότερο στη φύση των αρμοδιο... με την φύση των αρμοδιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Θα πρέπει να πούμε ότι... Α, να πούμε αυτό που είπε η Επιτροπή μας τελευταία θητεία, ότι ο συντονισμός των οικονομικών αρμοδιοτήτων θα πρέπει να θεωρηθεί ε, τμήμα μεικτών αρμοδιοτήτων και το άρθρο 136 μπορεί να υπερβεί αυτό το επίπεδο. Θα δούμε πώς θα φτάσουμε σε επιμερισμένες αρμοδιότητες στην οικονομική διακυβέρνηση. Έχουμε ήδη κάποια στοιχεία. Νομίζω ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπαίνει μόνο στο τέλος της διαδικασίας. Όταν θα έχουμε εντοπίσει τη φύση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στην ε, οικονομική πολιτική. Και αν πρέπει τέλος να γίνει μια αλλαγή της συνθήκης, η Επιτροπή μας είχε εγκρίνει μια έκθεση με διάφορες προτάσεις για μια αλλαγή της συνθήκης. Μπορούμε να επιλέξουμε να μην τις αναφέρουμε αυτές τις προτάσεις και να αναφέρουμε ε, αλλαγές που είναι πιθανές στα πλαίσια των σημερινών συνθήκων. Αλλά αν η Επιτροπή μας προτείνει αλλαγή των συνθήκων και υπάρχουν δυνατότητε, εγώ θα βλέπα πολύ πιο σημαντικές από αυτές που προτείνεται, ε, που τις έχουμε εγκρίνει ως Επιτροπή ΑΦΚΟ για, την, ε, για το μετασχηματισμό της οικονομικής πολιτικής και να είναι μεικτή αρμοδιότητα. Ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης, Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε εγκρίνει στο παρελθόν. Δεν νομίζω ότι αυτά που λέει η Σιλβή είναι τα πιο, οι πιο σημαντικές αλλαγές της συνθήκης. Γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ με εσά ότι αυτή η παράγραφος, η τελευταία δηλαδή, θα πρέπει να απαλληθεί. Ευχαριστώ Ρομπέρτο. σου. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό που η Επιτροπή ΑΦΚΟ εκδίδει μία γνωμοδότηση για την έκθεση που συντάσσουμε στην ΕΚΟΝ. Και χαίρομαι με τις προτάσεις ε, που θα κάνετε, που, κάνετε, εν Μην ξεχνάμε ότι εδώ θέλουμε να προσδιορίσουμε ποιε ιδέε τη Επιτροπή ΑΦΚΟ μπορούν να σωματωθούν στην ε, έκθεση τη ΕΚΟΝ. Καταρχά, το σχέδιό μου υποστηρίζει την ιδέα ότι οποιοδήποτε αναθεώρηση τη ε, οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύει την κοινοτική μέθοδο και όχι την διακυβερνητική μέθοδο. Σε πολλού τομεί ισχύει αυτό, αλλά ακόμα περισσότερο εδώ. Το σύνολο των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του τι είναι η οικονομική διακυβέρνηση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανοίξει τα μάτια της και το Κοινοβούλιο. Γιατί το Συμβούλιο, τέλο πάντων τα πράγματα είναι δεδομένα ε, με τη λειτουργία του Eurogroup. Αλλά παραδόξως το θεσμικό τρίγωνο, το μόνο όργανο που έφτασε στο τέλος αυτής της λογικής είμαστε εμείς. Αν θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε την κοινοτική μέθοδο θα πρέπει να τακτοποιήσουμε και τις ιδέες μας. Δεν θέλω να ξεκινήσω μια γενική συζήτηση εδώ, αλλά θέλω να μιλήσω λιγάκι τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεση που τελειώνω αυτές τις ώρες τώρα, υπάρχει ένα σημείο το οποίο αναφέρω και που νομίζω είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε μαζί με την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Είναι ο ρόλος και η θέση στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αυτή τη σύσταση για την ζώνη ευρώ, που είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει να μα εντοπίσει να ε, βλέπουμε τα διακυβεύματα, πώ μπορούμε να φτάσουμε σε μια σύγκληση στην ευρωζώνη. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι σε πιλωτική φάση για τις οικονομικές πολιτικές. Αλλά σήμερα δεν έχει ούτε νονό ούτε νονά. Αλλά τέλο πάντων νονά δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το μηχανισμό. Έχουμε μία εντύπωση ότι μεταξύ της Euro, του Eurogroup και της ε, Κομισιόν παίζεται ένα και ότι αυτό το έγγραφο δεν έχει την πραγματική σημασία που θα έπρεπε να έχει. Το να υπερασπιστούμε την οικονομική, την ε, κοινοτική μέθοδο, τι σημαίνει επίσης, να κάνει η Κομισιόν τη δουλειά της και να βρει ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της ε, μεθόδου. Για το δημοκρατικό έλλειμμα, συμφωνώ με τα ερωτηματικά που θέτεται για την λειτουργία τη διακοινοβουλευτικής διάσκεψης, αλλά η πραγματική προστιθέμενη αξία είναι ότι κάθε επίπεδο ελέγχου θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Και από αυτή την ε, σκοπιά, χου, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Στην έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είχα προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σύνομοθέτης για την ετήσια εξέταση της ε, ανάπτυξης. Αυτή η ετήσια εξέταση δεν είναι το πιο λειτουργικό έγγραφο, αλλά θα πρέπει ίσως να εξελιχθεί για να γίνει ένα πραγματικό πλαίσιο ε, διάγνωσης, για να δούμε ποιος είναι ο καταμερισμός των ρόλων, τι ρόλο παίζει το κάθε κράτος μέλος. Και θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς μπορεί να ενισχυθεί, να ενισχυθεί αυτός. Γιατί ε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαστε η κατάλληλοι το κατάλληλο βήμα για να γίνει αυτή η συζήτηση για την αξιολόγηση της κατάστασης. Σε σχέση τώρα με τις ε, προτάσεις του συναδέλφου Τζιγόν, ε, μία λέξη για την ευθύνη της Κομισιόν ε, στο εσωτερικό της Τρόικα. Εγώ είχα ακούσει μια δέσμευση του Γιούνκερ ότι θα τελειώσει η ιστορία της Γιούνκερ, της Τρόικα, και η ΕΚΤ ε, ουσιαστικά θα δολοφονεί στην Τρόικα μια και δεν θα έχει πια την δυνατότητα να συμμετάσχει. Τώρα, δύο σημεία, σύντομα. Και τα δύο συνδέονται με το θέμα της αναθεώρησης των συνθήκων. Εγώ φυσικά πιστεύω ότι αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ε, ΟΝΕ, κάποια στιγμή πρέπει να αναθεωρήσουμε τις συνθήκες. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις όμως για την ιδέα της ε, δικαστικοποίησης, της διαδικασίας για τα οικονομικά. Ένα πράγμα που δεν λειτουργεί στην Οικονομική Ομισματική Ένωση είναι υπερβολική, υπερβολικά πολλοί κανόνες που δεν γίνονται σεβαστοί. Και τα δύο είναι προβληματικά. Πολλοί κανόνες υπάρχουν και δεν γίνονται και σεβαστοί. Και το ένα μάλιστα επιφέρει το άλλο. Αν έχουμε πάρα πολλούς κανόνες και αν τους ε, δικασ ας πούμε, θα επιδεινώσουμε την κατάσταση. Γιατί αν δεν μπορεί να πει τίποτα το δικαστήριο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να είμαστε συνετοί. Παρότι θα πρέπει να στα κράτη-μέλη διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις να γίνονται με τη συμμετοχή και την ε, επιθυμία των κρατών μελών. Μεγαλύτερη συμμετοχή. Μπορούμε να δούμε το θέμα επίσης της ιεράρχησης το, των κοινωνικών δικαιωμάτων σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά και να δούμε τι έχει ε, προτεραιότητα. Αν δεν γίνει αυτό μέσω της ΟΝΕ, μπορούμε να δούμε ότι Τέλο πάντων, έχουμε την αναθεώρηση των συνθήκων, αλλά μπορεί να γι... μπορούμε να σκεφτούμε με διάφορους τρόπους. Τέλος πάντων, περιμένω όλες τις ιδέες από την ΑΦΚΟ ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και θα τις λάβω υπόψη μου γιατί, είναι, γιατί μας εμπλουτίζουν. Κοιτάξτε, Πρόεδρος, δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω το λόγο σε άλλους. Ο κύριος Κατρούκαλος και ο κύριος Λάινεν μου ζήτησαν το λόγο μόλις τώρα, αλλά ε, έχουμε πάρει ήδη πάρα πολύ χρόνο. Καταναλώσαμε και το χρόνο του κυρίου Πόνς, που δέχτηκε να μην συζητήσουμε το θέμα του σήμερα. Όμως θα συζητήσουμε την έκθεσή του 26 Φεβρουαρίου και θα υπάρχουν μόνο λίγες μέρες μετά για τις ε, τροπολογίες. Θα πρέπει να τις προετοιμάσετε από τώρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να παρακαλέσω τους κύριους Κατσρούγκαλο και Λάινεν να διεξαχθεί η συζήτηση, να παρέμβουν δηλαδή στη συζήτηση των τροπολογιών. Γιατί αλλιώς έχουμε κι άλλους που θα έρθουν τώρα. Να δώσω πάλι το λόγο στη Σιλβή και μετά να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σιλβή, ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδίω τους και τις συναδέλφους που ήταν παρόντες και παρούσες. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις απόψεις που θα ήταν πιο δίκαιο. Μία παρατήρηση. Η γνωμοδότησή μου εκδόθηκε πριν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα μην ερμηνεύουμε μέσα σε αυτήν κάποια ε, θέληση να μην τη λάβω υπόψη. Είναι γεγονός. Υπάρχει ισορροπία στο κείμενό μου, πιστεύω, και δεν νομίζω ότι πρέπει ο καθένας να βγάλει τα κερασάκια για να τα από το γλυκό. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία στο σύνολο. Για το θέμα βέβαια της αναθεώρησης των συνθήκων, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των συνθήκων για την οικονομική διακυβέρνηση. Αντιθέτως και ευχαριστώ την ε, Περβάνς για την αναφορά στο δικαστήριο. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να πάρουν δικαστικό χαρακτήρα οι αποφάσεις για το προϋπολογισμό. Όχι. Αλλά λείπουν δύο πράγματα που είναι χαρακτηριστικά των κρατών δικαίου. Η δυνατότητα να ζητείτε η ακύρωση των αποφάσεων και επίσης η δυνατότητα προσφυγής κατά μιας χώρας η οποία δεν σέβεται τις υποχρώσεις της. Δεν σημαίνει θα τη πούμε τι θα κάνει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα συζήτηση να γίνει πάνω σε μια αυστηρά λογική βάση. Για, όταν το δικαστήριο ακολουθεί τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, να μπορεί να τέμνει μια, ε, υπόθεση, σε μια υπόθεση, που ήταν για παράδειγμα η υπόθεση ε, ε, του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε το θέμα αυτό, βεβαίω λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, λεπτομέρειε τη εφαρμογή. όμως όμω υπάρχει στην κοινοτική μέθοδο, επί τη οποία όλοι ταχθήκατε, ένα τέτοιο μεγάλο κενό. Όμω η κοινοτική μέθοδο προβλέπει και δικαστήριο, που είναι αυτό το οποίο επιβάλλει το δίκαιο παραπάνω από τι χώρε μέλη. Βρίσκεται δηλαδή σε υπέρτερο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 28 Ιανουαρίου. Και στις 26 Φεβρουαρίου θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων και ε, στις 17 θα γίνει η ψηφοφορία. Και υπόσχομαι στους δύο συναδέλφους που δεν μίλησαν ε, σήμερα ότι θα μπορέσουν να παρέμβουν τις, ε, στις επόμενες συνεδριάσεις. Βεβαίως η Σιλβία αναμένει και τις δικές σας απόψεις. Ας περάσουμε τώρα στο θέμα υπαριθμών 6. Είχαμε συμφωνήσει ότι αναβάλουμε το θέμα του Εστεμπάν Γκονζάλες Πόντ. Ε, μόνο οι σοσιαλιστές έχουν διορίσει και ο που είναι ο, ο κύριος Σίλβα Περέιρα που θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον ε, κύριο Γκονζάλε Πόνς. Από τις άλλες πολιτικές ομάδες δεν έχουμε λάβει ακόμη τα ονόματα των σκιωδών εισηγητών. Θα ήθελα τώρα να έρθουμε στο υπαριθμό 7 της ημερησίας διατάξεως για το European Youth Event, Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νέων. Ε, να έρθουν εδώ κοντά μου οι συνάδελφοι. Ε, ε, συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για την μήνυ ακρόσια ό,τι αφορά το, ε, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τους Νέους που έλαβε χώρα τον περασμένο Μάιο στο Στρασβούργο με πολλούς ε, νέους που πρότειναν ιδέες στο Κοινοβούλιο. Σήμερα έχουμε προσκαλέσει τρεις νέους ε, έχετε τα βιογραφικά τους, γνωρίζετε από πού προέρχονται, τι αντιπροσωπεύουν. Ε, θα μας υποβάλουν έξι ερωτήσεις. Και έχουμε πολύ αυστηρούς ε, κανόνες γιατί οι γιατί νέοι αυτοί θα πρέπει να πάνε και σε άλλες επιτροπές, έχουν πολύ αυστηρό πρόγραμμα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Οι πρώτες ερωτήσεις θα είναι το πρώτο μπλοκ μάλλον ε, θα αφορά τις εκλογές. Ε, θα ακούσουμε τον ε, Μαντέα Μεχμούτ και την Λορεντάνα Ορτσίζα. Ποιος ξεκινάει? Μαντέα. So my, my, my Η πρώτη μου ιδέα είναι οι ηλεκτρονικές πληροφορίες. ως ε, πρόσθετο τρόπο έναντι της παραδοσιακής ψηφοφορία προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή ομάδων ε, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν καταφέρουν να συμμετάσχουν στις εκλογές και για ανθρώπους που ε, αμφιβάλλουν για το θέμα της ασφάλειας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το vd που είναι ένα σύστημα διπλής ασφάλειας το οποίο δίνει ε, και γραπτή απόδειξη ότι κάποιος ψήφισε ε, ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύει ε, και, το, και την ψήφο έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε επαληθεύσεις εκ των υστέρων. οι συζητήσεις μεταξύ νέων στην Ευρώπη δείχνουν ότι τίθεται θέμα ενοποιημένου συστήματος ψηφοφορία. Ίσως θα έπρεπε να μειωθεί ε, το ηλικιακό όριο στα 16. Ε, το δικαίωμα ψηφοφορία είναι σημείο κλειδί της δημοκρατικής ε, συμμετοχικής διαδικασίας. Και το δικαίωμα ε, του εκλέγει και του εκλέγεστε είναι επίσης κέριο δικαίωμα. Δεν έχει νόημα να έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ε, στα εκλογικά του συστήματα. Η Αυστρία και η Μάλτα χρησιμοποιούν το όριο των 16 ετών, ε, για παράδειγμα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ε, δημοκρατική πρόκληση και δημογραφική πρόκληση. Κάθε χρόνο ο αριθμός των νέων μειώνεται. Ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος αριθμός των δημοκρατικών χωρών βλέπουν ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων μειώνεται. Γι' αυτό το λόγο οι πολιτικές συζητήσεις μπαίνουν στο περιθώριο, κάτι που δημιουργεί δημοκρατικό έλλειμμα. Για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η νομοποίηση των πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει περισσότεροι νέοι να ψηφίζουν και να συμμετέχουν. Αυτό μπορεί να γίνει με την μείωση του ορίου στα 16 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργούσε και ένα πιο ενοποιημένο εκλογικό σύστημα είναι ένα θέμα το οποίο οι νέοι το συζητούν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ Λορεντάνα. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να απαντήσουν. Τζο Λάινεν. Έχουμε ήδη τρεις συναδέλφους. Yeah, uh, one minute λεπτό καθένας. Ούτε ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πρόταση. Ε, θα θέλαμε πράγματι ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα, ένα ενιαίο σύστημα ψηφοφορίας. Χωρίς μικρόφωνο μιλτής δυστυχώς. Oh, yeah, yeah, You see, the next will be the alarm clock ringing that we have to go out of the room. <laughs> Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι ο συναγερμός που πρέπει να εκενώσουμε την αίθουσα. Ε, λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε που αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σύστημα. Υπάρχουν πράγματι πολλές αδυναμίες και η Επιτροπή μας ακριβώς εργάζεται επί αυτού του θέματος και ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας θα, θα καταφέρουμε να κάνουμε μια πρόταση για τις επόμενες ευρωεκλογέ του 19. Οι πρόεδρος και εγώ είμαστε ε, αυτοί που, γνωμοδο... που έχουν αναλάβει την έκθεση για αυτό το ζήτημα. Ε, θα πρέπει οι ευρωπαϊκές εκλογές να είναι πιο ελκυστικές. Ευχαριστώ πολύ για τη σκέψη σας. Uh, thank you, Richard Corbett. Richard Corbett. Θα μπορούσατε να συστήνετε κιόλα στους συναδέλφους. Εκπροσωπείτε τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ονομάζομαι είναι Richard Corbett από το Εργατικό Κόμμα, ε, μέλος των σοσιαλιστών. Ε, συμμετείχα στην, ε, την εκδήλωση αυτή στο Στρασβούργο τον περασμένο Μάιο. Ε, Παντεσία απόψεων, συζητήσεων. Ε, ήταν πολύ ωραίο να δούμε τόσους ε, νέους, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ο χρόνος είναι περισμένος. Συνεπώς θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα του συστήματος ψηφοφορία. Και στην αρχή, αν δούμε ότι είναι, αν πούμε ότι είναι αρχή, ε, ότι το όριο ε, για να ψηφίζει κάποιο νέο θα πρέπει να είναι τα 16 χρόνια. Το υποστηρίζω. Το Εργατικό Κόμμα στην Βρετανία επίση το στηρίζει. Και αν κερδίσουμε το Μάιο τι ε, κοινοβουλευτικέ εκλογέ μα θα προσπαθήσουμε να περάσουμε νόμο που να κατεβάζει το όριο στα 16. Ευχαριστώ. Είμαι ο George Σέπφλιν από το ΕΛΚ της Ουγγαρίας. Δύο σχόλια. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κοιτάξτε το παράδειγμα την εμπειρία της Εστονίας. Ε, εκεί ε, εφαρμόζεται ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ε, δεν είναι ότι δεν έχει προβλήματα. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα αν κάποιος το προσπαθήσει. Και ίσως κάποιες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες. Μετά, τη μείωση του ορίου στα 16. δεν έχω πρόβλημα με αυτή, καθ' αυτή την πρόταση. Να πω όμως το εξής. το κέντρο της δημογραφικής βαρύτητας στην Ευρώπη αυξάνεται. Πολύ σύντομα, 50-60% του πληθυσμού θα είναι πάνω των 65 ετών. Θα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, ε, θα ζουν μέχρι τα 125 τους, ενδεχομένως εσείς οι ίδιοι. Οπότε ίσως θα έπρεπε να εστιάσουμε στους άνω των 65 όχι στους κάτω των 18. Αυτό είναι το πιο λογικό. Ε, και η μείωση των, ε, της συμμετοχής προς τα εκεί θα έπρεπε να μας ε, κατευθύνει. Ε, ίσως θα πρέπει να δούμε την ε, διεύρυνση των ε, ευρωπαϊκών δημογραφικών στοιχείων και ενδεχομένως ένα δημοψήφισμα επί αυτού θα ήταν καλό. Ωραία. Άλλη μία παρέμβαση, ο κ. Σόλτς. Από την Γκουε. E. Έχουμε δύο παρατηρήσεις. Είμαστε υπέρ του όλη των 16 ετών. Ε, ασφαλώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλη την κοινωνία, αλλά η, δυνατότητα των νέων να συμμετάσχουν και να επηρεάσουν την πολιτική είναι πολύ σημαντική. Ε, θα έπρεπε να έχουν το δικαίωμα ε, να επηρεάζουν την πολιτική μας. Μετά, η μείωση της συμμετοχής σε εκλογές δεν οφείλεται στο ίδιο το σύστημα ε, μόνο. Α, οφείλεται και στην έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης ε, από πλευρά των νέων και γενικότερα από πλευρά των εκλογέων των ψηφοφόρων ε, στην δυνατότητα του συστήματος, του ευρωπαϊκού συστήματος να δώσει λύσεις. Και θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούνται πολιτικές οι οποίες να μπορούν να κατανοηθούν από τους πολίτες έτσι ώστε να τους οθήσουν να συμμετάσχουν σε εκλογές και να ψηφίζουν. Ωραία. 1,5 λεπτό 1,5 λεπτό σε καθένα από του συναδέλφου Λορεντάνα και Μαντέχα. Δεν, μπορείτε, δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε με όσα ακούστηκαν. Μπορείτε να απαντήσετε απλώ. Uh, you ε, ευχαριστώ. Ναι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για, που εξηγούν την αποχή. Το εκλογικό σύστημα είναι ένας από αυτού. Υπάρχουν άνθρωποι που ε, σπουδάζουν στο εξωτερικό, για παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιοι ε, με, άνθρωποι με αναπηρίε ε, σωματικέ ή πνευματικέ. Και ε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορούσε να του συμπεριλάβει, να του δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν και αυτοί. Ασφαλώ υπάρχουν πολλά προβλήματα ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ένα διπλό σύστημα επαλήθευση. Υπάρχουν και άλλε δυνατότητε. Ξέρω ότι Υπάρχουν ε, σίγουρα χώρες που θα προσπαθήσουν να μας χακάρουν, αλλά ε, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και να αυξάνουμε σιγά σιγά την ασφάλεια. Ε, να μην πούμε δηλαδή ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι δεν θα το εισάγουμε ποτέ. Ε, οι νέοι του Ηνωμένου Βασιλείου σίγουρα θα ακούσουμε πολύ χαρά αυτό που είπατε γιατί το έχουμε διεκδικήσει. Έχουμε διεκδικήσει τη μείωση του ορίου. Ε, του ηλικιακού ορίου. Ε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν θα είναι ίσως ε, έτοιμοι και όριμοι ε, στα 16, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε παράλληλα με κάτι άλλο, με την εφαρμογή ε, του, με την εισαγωγή του ως υποχρεωτικού του μαθήματος στις ε, συνείδησης πολίτη ε, στα σχολεία. Θα ήταν κάτι ενδιαφέρον αυτό ο συνδυασμό των δύο έτσι ώστε είναι να αποκτήσουν φωνή. Ευχαριστώ. Ωραία. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα. Θα σας ξαναδώσω το λόγο για το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας. Your, your interest, um, you can go broader, of course. Yes, you're welcome. Thank you. Um, the next team. Ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των νέων, στο Στρασβούργο ε, Είχαμε συζητήσει το θέμα του αν χρειάζονται ποσοστώσεις ή όχι. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζονται ποσοστώσεις για τους νέους, υπέρ των νέων. Ε, η συμμετοχή των νέων ε, θα μπορούσε να ε, υποστηριχθεί αν εκλέγαμε έναν σύμβουλο, νέο σύμβουλο από κάθε χώρα, 28. Ε, ε, εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα, μπορούσαν, θα μπορούσε ένας από αυτούς να συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ παράλληλα με εσά να σας συμβουλεύει από την πλευρά των νέων μια, ε, ένας, ε, μια θέση, αμοιβόμενη θέση εργασίας αυτά τα άτομα, οι σύμβουλοι θα είναι σε επαφή με τις οργανώσεις των νέων στις χώρες τους και ταυτόχρονα θα παρακολουθούν το τι ακριβώς κάνετε εδώ και θα συμμετέχουν όχι μόνο ως παρατηρητές αλλά και ως ενεργά μέλη των επιτροπών. Ε, θα πρέπει να, να ζητάει τη γνώμη των πολιτών πιο συχνά για τα διάφορα θέματα, με δημοψηφίσματα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει όλοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη γνώμη τους, να παρουσιάζουν τη γνώμη τους, ιδιαίτερα αν δεν είναι μέλος κάποια, μέλη κάποιας ένωσης συνδικάτου κλπ. Η συμμετοχική δημοκρατία θα πρέπει να αναγνωριστεί από όλου τους πολίτες μας, προκειμένου αυτή να είναι ε, να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες. Η συμμετοχική δημοκρατία μπορεί να πετύχει μόνο αν πληρούνται δύο όροι. Πρώτον, η όλη διαδικασία είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και δεύτερον, έτσι, να είναι διαρθρωμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η συμμετοχή του κοινού να έχει αποτέλεσμα, πρακτικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει το πλαίσιο να μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις ανάγκες των πολιτών, και να γίνεται πρώτα μια διαβούλευση προκειμένου να συζητώνται οι διάφορες ιδέες για κάθε πρόβλημα. Ο άμεσος διάλογος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα και παντού έτσι ώστε οι νέοι να συμμετάσχουν. Ε, τα δημοψηφίσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό βήμα για να, για να βελτιώσουμε τη συμμετοχική δημοκρατία. Και όπως είπα, κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Uh, we already have Bresso who like to ask the questions and George and... Η κυρία Μπρέσο θέλει να κάνει ερωτήσεις, ο Γιώργος Κατρούγκαλος επίσης. Ευχαριστώ. Βάλτε σας παρακαλώ τα ακουστικά σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις για το θέμα του Συμβούλου Νεότητας γιατί νομίζω ότι η μείωση του δικαιώματος ψήφου στα 16, με το οποίο συμφωνώ, θα σήμαινε ότι και πιο νέοι θα εκλέγονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ούτως ή άλλως έχουμε ήδη νέους οι οποίοι μπορούν να εκπροσωπήσουν και τα συμφέροντά σας. Μπορεί να υπάρχουν ε, και λομπίστε πληρωμένοι από το Κοινοβούλιο για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά σα. δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Ε, αντίθετα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του δημοψηφίσματος. Προτείνεται ένα δημοψήφισμα συμβουλευτικού χαρακτήρα για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν. Προφανώς, το θέμα του δημοψηφίσματο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα πανευρωπαϊκό, α πούμε, δημοψήφισμα θα ήταν η λύση για να ξεπεράσουμε και τα εθνικά δημοψηφίσματα για την τροποποίηση των συνθήκων, Φερρυπίν. Ένα μεγάλο δηλαδή ευρωπαϊκό δημοψήφισμα για την τροποποίηση των συνθήκων και θα έδινε και νόημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς αυτό το δημοψήφισμα το έχετε φανταστεί επί επιμέρου σημείων ή το θεωρείτε ω ένα εργαλείο α πούμε για να ψηφίσουμε και έναν εκλογικό ας πούμε νόμο ενιαίο για όλε τι χώρε ή ένα πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα για να αποφασίσουμε για την τροποποίηση των συνθήκων. Ευχαριστώ Γιώργος. Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας και που ήρθατε. Ε, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι η νέα γενιά είναι απομακρυσμένη από την πολιτική. Όχι μόνο οι νέοι δηλαδή, και λιγότερο νέοι. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε παραδοσιακές μορφές ε, δημοκρατίας μαζί με την άμεση δημοκρατία για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στην πολιτική σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, ευρωπαϊκό κτλ. Για την πρότασή σας για το πανευρωπαϊκό ρεφερέντουμ, ιδέα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή για το πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα. Γιατί μου αρέσει αυτή η ιδέα της άμεσης δημοκρατίας και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό δήμο, δεν είναι επιθυμητό ούτε δυνατό. Αλλά μπορούμε να έχουμε κοινέ συζητήσει γύρω από ένα κοινό θέμα. Να έχουμε λοιπόν ένα οργανωμένο δημόσιο χώρο που είναι προϋπόθεση για να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις. Επίσης, μία ιδέα που έχει δοκιμαστεί όταν οι Ισλανδοί συνέτασαν το νέο του σύνταγμα είναι η συμμετοχή των κοινωνικών μέσων στην πολιτική συζήτηση. Όταν η συνέλευσή τους έφτιαχνε το νέο σύνταγμα, ε, φόρτωναν την νομοθετική δουλειά τους κάθε μέρα στο ίντερνετ και παίρναν ιδέες από τα μέσα, από τα κοινωνικά μέσα. Δεν είμαστε όλοι τόσο ενημερωμένοι με τις νέες τεχνολογίες όσο εσείς, αλλά νομίζω ότι το να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες στο δημόσιο βίο θα ήταν χρήσιμο. Εμείς δεν είμαστε τόσο πειθαρχημένοι στον χρόνο, βλέπετε αγαπητοί νέοι όσο εσείς. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Συμφωνώ να μειώσουμε το όριο ηλικία για την συμμετοχή στι εκλογέ στα 16. Είναι πολύ σημαντικό για την συμμετοχή των νέων και στην Καταλωνία το δεχτήκαμε αυτό στι 9 Νοεμβρίου. Ψήφισαν και οι νέοι, δηλαδή λιγότερο νέοι, οι πιο νέοι για τα δημοψηφίσματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δημοψηφίσματα για πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Και καθιστά όχι μόνο δυνατό τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, αλλά και εύκολη και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά από όλα τα κράτη-μέλη, να χρησιμοποιούν λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη την τεχνολογία για αυτό το σκοπό για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή και η δημοκρατία γίνονται πράγματα πάρα πολύ εύκολα και πλησιάζουμε ακόμα περισσότερους πολίτες. Ευχαριστώ που ήρθατε επίσης. Ευχαριστώ. Ο Σύμβουλος Νέων. Μου φαίνει στο μυαλό ορισμένε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Πρώτα, ξεκινάτε από την υπόθεση ότι είναι ομοιογενή η προσδοκίε, φιλοδοξίε των νέων. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεύτερο, θα πρέπει να εκλέγεται αυτός από κάθε συγκεκριμένη χώρα. Μάλιστα. Και τρίτο, εκλεγμένο εκπρόσωπο ή σύμβουλο νέων θα έχει πολύ διαφορετικά καθήκοντα αν είναι για παράδειγμα Γερμανός ή Μαλτέζος ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των προσώπων που τον εκλέγουν. Τέλο, δεν είμαι αντίθετο βέβαια με την αρχή του ε, Συμβούλου των Νέων τότε όμως μπορεί και άλλες ομάδες να θέλουν να έχουν πρόσωπο ή σύμβουλο. Όπως για παράδειγμα οι άνθρωποι με ανάγκες. Να δούμε λοιπόν τι είδους ομάδες θέλουμε να εκπροσωπούνται. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Εσείς τώρα έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ναι, θα είναι εκλεγμένοι στις χώρες τους και σε ένα ιδιώδη κόσμο θα έχουμε τον ίδιο αριθμό συμβούλων όπως και ευρωβουλευτών. Γι' αυτό ε, λέμε να υπάρχει, να υπάρχει ε, εισαριθμία. Θα είναι δύσκολη δουλειά του προσώπου αυτού, αλλά τουλάχιστον θα έχει φωνή και άμεση επαφή με τους ευρωβουλευτές. Για την ώρα, αν είμαστε τυχερές, στέλνουμε ένα tweet και απαντάτε, αν είμαστε τυχεροί. Αν είμαστε τυχερές, επίσης, μπορούμε να έρθουμε να σας μιλήσουμε για δύο λεπτά. Ενώ εκεί θα υπάρχει μια σταθερή επαφή. Θα μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για το τι ενδεχόμενα να πείτε εσείς στη συναντήση σας. Βέβαια φαίνεται φιλόδοξο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Σας ευχαριστώ. Okay, so to answer the question, yeah, I think the... Για να απαντήσω στην ερώτηση ναι, ε, αυτά τα δημοψηφίσματα θα πρέπει να είναι εργαλείο και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν θα καλούμαστε να λάβουμε πολύ μεγάλη σημασία στις αποφάσεις. Και ναι, θα, ε, πρέπει να γίνει ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρο και εμεί να συμβάλλουμε στη δημιουργία του. Οι πολίτες από όλη την Ευρώπη εκεί να μπορούν να συνδιαλέγονται και να εκφράζουν απόψεις. Και χαίρομαι που βάλατε και το θέμα των κοινωνικών μέσων, γιατί εμείς είμαστε βέβαια πολύ κοντά σε όλα αυτά τα εργαλεία. Και μάλιστα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νέων αυτό ήταν το βασικό κανάλι επικοινωνίας μας γιατί εκεί εκφράζουμε τις απόψεις μας και τα όσα θέλουμε. Πάντως ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε εδώ γιατί αυτό είναι το είδος συμμετοχικής δημοκρατίας που φανταζόμαστε και θέλουμε να την ενισχύσουμε και σε κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό κλπ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τώρα δύο ε, γυναίκες που έθεσαν ερωτήσει. Τώρα έχουμε και έναν άντρα που έχει και αυτό το δικαίωμα. Α, να κάνει μάλιστα το διπλό αριθμό ερωτήσεων. Μιχαήλ Μάιερ, λοιπόν, δύο ερωτήσει. Ευχαριστώ. Πρώτα να πω ότι είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μένα που με προσκαλέσατε εδώ για λογαριασμό παραπάνω από 5.000 νέων 5.000 νέων που ε, συναντήθηκαν στην εκδήλωση ε, νεολαία. Είναι σπουδαία υπόθεση που με προσκαλέσατε εδώ. Θέλω να μιλήσω για τα όργανα και τι διαδικασίες. Αλλά αυτά όλα συγχωνεύονται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, και το πιο σημαντικό νομίζω, είναι να δοθούν περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα να δώσετε απλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα ανάληψη πρωτοβουλία απλώ. Από τα πιο μεγάλα κοινοβούλια στον κόσμο που εκλέγεστε από πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδε εκατομμύρια ανθρώπων ε, και από 28 χώρε μέλη και είναι το μόνο κοινοβούλιο που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον που δεν έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Να του δοθεί λοιπόν αυτό το δικαίωμα. Δεύτερο, το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω υπάρχει η συνθήκη τη Λισαβόνα, οι συνθήκε τη Ρώμη κτλ. Όπω λέγονται όλε αυτέ οι συνθήκε τέλο πάντων. Μπορείτε να κάνετε 20 συνθήκε και να δώσετε σε κάθε μια από αυτέ το όνομα μια πρωτεύουσα. Αλλά αυτή η συνθήκη τη ε, Λισαβόνα, δύσκολο, να, αδύνατο να την κατανοήσει ο απλό άνθρωπο. Οι νέοι λοιπόν και εγώ, στο όνομά του, ε, θα ζητήσουμε να φτιάξετε ένα απλό, ευνόητο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου να μπορεί να βασίζεται ο κάθε πολίτης. Αυτό θα βοηθήσει τον κόσμο και να ταυτιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις αξίες που εκφράζει. Αναλογιστείτε το Σύνταγμα των Ενωμένων Πολιτειών, που είναι εύκολο να το κατανοήσει ο καθένας. ο χάρτης των δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να είσαστε ε, επιχειρηματίας ή νομικός ότι αν δεν έχετε υπόψη σας όλες τις ε, συνθήκες πάνω σε οποίες στηρίζετε δεν μπορείτε να το διαβάσετε. Να δώσετε λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα. Περισσότερε εξουσίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα πρωτοβουλία και να φτιάξετε ένα σύνταγμα που να μπορεί να το καταλάβει ο κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Χαουρέγγι. Θα ήθελα να παρουσιάσω στους νέους μας την εξής ε, σκέψη. Πολλά από όσα ζητάτε απαιτούν ε, ευρωπαϊκές ε, χώρες να εκχωρήσουν εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αν θέλουμε ένας ευρωπαϊκός νόμος να επιτρέπει την ψήφο στα 16, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια τέτοια νομοθεσία. Άλλο παράδειγμα, για να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Σύστημα να το προβλέπει για να ε, εισαχθεί ένα κοινό μάθημα για την Ευρώπη στα ευρωπαϊκά σχολεία θα πρέπει επίσης τα εθνικά εκπαιδευτικά σύστημα να προβλέπουν τη δυνατότητα αυτή. Οπότε η σκέψη μου είναι η εξής. Όλα όσα ζητάτε απαιτούν ε, μια κινητοποίηση υπέρ της περισσότερης Ευρώπης για να πετύχουμε την καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ Ραμόνο Τζο Λάινεν. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη της Ένωσης από το 1984. 30 χρόνια. αρχαίος πινέδι. Στόχος σημαντικός. Ως τώρα δεν κατόρθωσαμε να τον επιβάλλουμε. Οι συνθήκε είναι πολύ περίπλοκε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη βάση. Εμεί το ονομάσαμε αυτό συνταγματικό ε, κείμενο τη Ένωση, γιατί όταν λέει κανεί σύνταγμα πολλοί φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να γίνει ένα υπερκράτο. Όμω όπω είπατε ένα κείμενο που να το καταλάβει κανεί. Αυτό όμω που μπορεί να καταλάβει κανεί είναι ο χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων. Εγώ μάλιστα λέω να το διαβάσετε όλοι στα σχολεία. Εκεί είναι εκφρασμένες οι αξίες της Ευρώπης στις οποίες θεμελιώνονται πάνω τα θεμελιώδη δικαιώματα με τη σειρά τους. Αυτό το τμήμα των συνθήκων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω πρώτο και δεύτερο μέρος κάποια στιγμή να μπορέσουν να περιοριστούν, αν το θέλετε έτσι, να συρρυγνωθούν σε ένα ενίο κείμενο το οποίο να μπορούν να κατανοήσουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μάιτε Ρουίση. Όπως, το είπε και, όπως είπε και ο Ραμόν Χάουραγη, πράγματι ορισμένα από αυτά που διεκδικείται και τα οποία είναι πολύ ε, θετικά έχουν σχέση με την εκόρση αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την οικοδόμηση της ε, μαθύτερης Ευρώπης. Ε, πιστεύω ότι χρειάζεται απαραίτητος ένα μάθημα για την Ευρώπη στα σχολεία γιατί το να προωθούμε τις ευρωπαϊκές και δημοκρατικές αρχές ε, από πολύ μικρή ηλικία θα μας ε, βοηθούσε στο να αποφύγουμε την ριζοσπαστικοποίηση των παιδιών και ε, να καταπολεμήσουμε τη βαρβαρότητα. Χρειάζεται όμως κάτι τέτοιο τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος, δημοκρατικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Ε, νομίζω ότι όσα είπες ε, είναι πραγματικά υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Είναι σαν να ε, είσαι εγγονός του Σπινέλη. Σε 20-30 χρόνια όλα αυτά που ζητάς πιστεύω ότι ε, θα είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό παρόλο που σήμερα μπορεί να φαίνονται ε, παράξενα αυτά που ζητάς ε, σήμερα. Νομίζω και ελπίζω ότι θα προωθηθούν. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρέσο. Ευχαριστώ πολύ για την ιδέα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Θα δουλέψουμε σε αυτό το θέμα και ελπίζουμε θα τα καταφέρουμε. Γνωρίζετε ότι υπάρχει η ομάδα Σπινέλη. Θα μπορούσατε να ζητήσετε μια επαφή με αυτή την ομάδα έτσι ώστε το θέμα να συζητηθεί βαθύτερα. Ε, σας προσκαλώ να το κάνετε και ταυτόχρονα σας ευχαριστώ για αυτό τον ε, ε, ε, φιλοευρωπαϊκό αέρα που φέρατε εδώ μέρος των νέων. Μακάρι και οι υπόλοιποι να ήταν όλοι σαν και εσά. χωσέ Μαρία Παρακαλώ εξακολουθήστε να διακρικείτε, να ζητάτε, να επικρίνετε γιατί η Ευρώπη ε, κινείται με ταχύτητα χελώνας. Ελέφαντα θα έλεγα. Η συνάδελφος ε, είπε ότι σε 20-30 χρόνια αυτά θα είναι πραγματικότητα. Εγώ θα ήθελα όλα να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα γιατί τότε δεν θα ζω πιθανότατα. Θα ήθελα σε 5, σε 10 χρόνια να τα έχουμε πετύχει. Είστε νέοι αλλά είστε ισχυροί οπότε παρακαλώ συνεχίστε να ζητάτε, να απαιτείτε, να προκαλείτε. Ευχαριστώ. Uh, thank Σας ευχαριστώ για τις αντιδράσεις σας. Να απαντήσω αν με επιτρέπετε σύντομα. Να πω ότι όλες οι ιδέες που υποβάλλουμε χρειάζονται περισσότερη συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για εκχώρηση κυριαρχίας των χωρών μελών υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πάει και στην Κίνα και στο Καζακστάν πριν από λίγους μήνες και για πρώτη φορά στη ζωή μου πέρασα από σύνορα. Χρειάστηκε να περιμένω στα σύνορα, να με ψάξουν τα τελωνία κτλ. Οι γονεί μου είπαν ότι προ 25 ετών, όταν από την Αστρία ήθελαν να πάνε στην Ουγγαρία να ψωνίσουν, σχεδόν διέλυσαν το αυτοκίνητο οι τελωνοφύλακε για να βρουν ενδεχομένως ε, λαθρέα τσιγάρα ή ενόπνευμα κτλ. Έτσι λοιπόν η γενιά μου έχει μεγαλώσει μέσα σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, σε μια Ευρώπη συνδεδεμένη, με ένα ενίο νόμισμα οι περισσότεροι από μας. Αυτό που βρίσκουμε εμείς είναι ότι η Ευρώπη κινείται αργά, σαν ελέφαντας τόσο αργά, αλλά κινείται παρόλα αυτά. Νομίζω ότι χρειάζεται να θέτετε θέματα, έστω και αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν αύριο, αλλά να εκφράζετε τις επιθυμίες αυτές και γι' αυτό σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Με μια φράση, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, ακούσατε από τους συναδέλφους μου ότι εκτιμούν αυτή την ανάσα φρέσκο αέρα που φέρατε εδώ και τις ε, ε, προτάσεις σας. Νομίζω οι περισσότεροι όμως από εμά θαύμασαν αυτή την δέσμευση που έχετε για την Ευρώπη. Και ελπίζουμε ότι Θα αντιληφθείτε κι εσείς βέβαια ότι η Ευρώπη δεν είναι μοναχά δικαιώματα και καταρρύψει των συνόρων κτλ. Αλλά είναι και υποχρεώσεις. Πολλοί από εμά που σας βλέπουμε ως εκπροσώπους της νέας γενιάς ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα σας παραδώσουμε τη σκητάλη και εσείς θα αναλάβετε πλέον από εκεί και πέρα την ευθύνη για τη λειτουργία της Ευρώπης και ότι επομένω στα χέρια σας η Ευρώπη θα είναι ασφαλής. Σας, ευχα... σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Συνεχίστε με την ε, ε, δέσμευσή σας και κολλήστε και άλλους ε, το μικρόβιο αυτό και σε άλλους νέους. Ευχαριστώ πολύ.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 Dear colleagues, can we just, Mercedes? The Italians are not very disciplined, I must. Again. Yeah. Okay. Could we, could we just... Ε, θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε ένθερμα ε, ε, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει δείξει πολύ γενοδορία κατά τη διάρκεια της Ιταλικής ε, Προεδρίας, μας ενημέρωσε ε, για την, το έργο της Προεδρίας. Ε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε ξανά μαζί μας για να μας παρουσιάσετε τα συμπεράσματα από το εξάμεινο της Ιταλικής Προεδρίας. Παρακαλώ σας δίνω το λόγο. Of course, thank you for, for the invitation. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν εδώ τον Ιούλιο και κατά τις υποσχέσει μου. Είχα πει θα ξανάρθω για να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα της ιταλική Προεδρίας και τις προκλήσεις που μας περιμένουν. Θα είμαι σύντομο, ούτω ώστε να έχουμε το χρόνο για όσους από εσά μπορούν να παραστούν να μπούμε σε συζήτηση. Ξέρετε ότι για μας η Προεδρία ήταν οι πρώτοι έξι μήνες μιας πενταετούς αλλαγής. Ξέραμε ότι το εξάμεινό μας θα ήταν ένα ατυχές εξάμεινο. Ήμασταν ε, στην Προεδρία τον Αύγουστο και ήμασταν στην αρχή μιας ε, θεσμικής μετάβασης. Και τελικά πήγε ομαλά το πράγμα, αλλά δεν ήταν καθόλου δεδομένο σίγουρο στην αρχή. Καταφέραμε με τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Φανρομπάη και σας να διαχειριστούμε μια ομαλή μετάβαση και να πάμε σε ένα σημείο πρωτοφανές και χωρίς επιστροφή. Την ε, αποκοινού επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμείς μαζί με άλλες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο και χάρη σε εσά και χάρη στην ομοφωνία των πολιτικών σας ομάδων είπαμε ότι θα πρέπει ε, η επιλογή αυτή να έχει και μια πολιτική βάση. Σεβαστήκαμε νομίζω τη θέληση των ε, Ευρωπαίων πολιτών διορίζοντας τον ε, Jean-Claude Juncker και φτάσαμε σε αυτό το σημείο χωρίς επιστροφή. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο της συνθήκης, εφαρμόσαμε αυτό το σημείο της συνθήκης αλλά για να το παγιώσουμε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά σε αυτή τη θητεία. Έχουμε λοιπόν, ε, είχαμε αυτούς τους έξι μήνες που προεδρεύσαμε σε ένα νέο πολιτικό κύκλο και όπου η έμφαση και η εστίαση ε, ήταν στην ανάπτυξη και στην ευελιξία. Είμαστε ικανοποιημένοι με τα πρώτα βήματα που σημειώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον πρόεδρο Γιούνκερ και πιστεύουμε ότι ήταν σημαντικό που μας παρουσίασε τις δύο βασικές προτάσεις, το σχέδιο για τις επενδύσεις, παρότι μπορεί να πιστεύετε ότι έχει αδύναμα σημεία, ε, η διαδικασία είναι διαδικασία στην απόφαση. Θα δουλέψουμε κι εμείς και εσείς από τη πλευρά σας, εμείς ως Ιταλία στο Συμβούλιο Υπουργών, αλλά και εσείς μαζί μας. Και είναι σημαντικό ότι λέμε ότι η αρχή είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Να ε, κινητοποιήσουμε την υπάρχουσα ρευστότητα, ε, προς, την, προς το κοινό καλό, ας πούμε, με έργα για το κοινό καλό. Και ήταν μία από τις προτεραιότητες στο πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στις 2 Ιουλίου στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό. Νομίζουμε ότι μέσα από τις ισχύουσες συνθήκες μπορούμε με πιο φιλικό τρόπο να εφαρμόσουμε τους ισχύοντες οικονομικούς κανόνες, αλλά με, έχοντας κατά νου την ανάπτυξη. Έχουμε αυτή την ανακοίνωση για την ευελιξία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι το πρώτο βήμα αυτής της προσπάθειας. Παρότι, κατά την άποψή μας, υπάρχει το περιθώριο ευελιξίας για να προωθήσουμε την ευελιξία και να βάλουμε την ευελιξία στην υπηρεσία μιας νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Για μας, ε, πολιτικά, πολιτικός οι δύο προτάσεις τη Κομισιόν είναι πολύ σημαντικέ. Η πρώτη για τι επενδύσει, η δεύτερη για την ευελιξία. Το δεύτερο βασικό κεφάλαιο του εξαμήνου της Ιταλικής Προεδρίας ήταν να σπρώξουμε το Συμβούλιο να είναι πιο συνεπές ε, και πιο σαφές σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρετε ότι πρέπει να καλύψουμε ένα κενό ανά, ανάμεσα στην τακτική διαδικασία επί και το ρόλο, τον κλασικό ρόλο ως θεματοφύλακα ε, των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το νέο άρθρο 7 της συνθήκης. Θα πρέπει εσείς στο Κοινοβούλιο να κάνετε τη ε, συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο πάντα αρνιότανε να κάνει αυτή τη συζήτηση, να προωθήσει, να επιτρέψει αυτή τη συζήτηση. Το αποτέλεσμα που πετύχαμε και η πολιτική δέσμευση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων είναι να γίνει τακτική συζήτηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το κράτος δικαίου, για τις ε, δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι μία ακόμα απάντηση σε αυτή την έκκληση για αλλαγή που ε, διατύπωσαν οι πολίτες μας στις ευρωπαϊκές εκλογές και που σας έφεραν σε αυτό το θόκο εδώ. Όχι μόνο να έχουμε λοιπόν μία τακτική συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία φορά το χρόνο, αλλά να το κάνουμε πέραν αυτή της μίας ε, θεσμοθετημένης φοράς και όποτε είναι απαραίτητο. βάζουμε έμφαση στο δυναμικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και να προωθήσει την ασφάλεια. Βάζουμε επίσης έμφαση στο σεβασμό του κράτους δικαίου, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε την απειλή της τρομοκρατίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν σκεφτόμαστε ας πούμε πώς θα συμφωνήσουμε για την οδηγία PNR και πώς θα τροποποιήσουμε τη Συμφωνία Σέγγεν για να διευκολύνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά θέτουμε παρόλα αυτά έμφαση στα νέα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να προωθήσουμε την ασφάλεια. Βάζουμε λοιπόν έμφαση και στο θέμα του κράτους δικαίου. Είναι ένα άλλο ε, στοιχείο το οποίο πρέπει να αντισταθμίσουμε. Δηλαδή από τη μία το δικαίωμα στην ασφάλεια και από την άλλη τα θεμελιώδη δικαιώματά μας εντός Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτά τα σταθμίζουμε. Κάτι άλλο, κάτι άλλο που συζητήσαμε λεπτομερώς με το Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς. Και που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμείναμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, να κάνουμε μια αναθεώρηση για τον τρόπο με τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λειτουργούν σήμερα στα πλαίσια των ισχυουσών συνθήκων και δεύτερον να επανεκκινήσει η συζήτηση και η δράση που προωθήθηκε από την έκθεση για την οικονομική διακυβέρνηση. Η Προεδρία είναι κυλιόμενη, όπως ξέρετε. Ως μέλος της Ιταλικής κυβέρνησης και ως Ιταλία θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι, γιατί ήδη έχουμε θέσει επιτάπητο το θέμα του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα θέλαμε να κάνουμε αυτό που κάνετε εσείς σε αυτή την Επιτροπή, Πρόεδρε, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, κάνετε μία διπλή προσπάθεια. Τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και καλύτερα εντός των υπαρχουσών συνθήκων, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό των σημερινών συνθήκων και πώς μπορούμε να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα για το εγγύς μέλλον, που για μένα εγγύς μέλλον σημαίνει πριν το 2019. Ίσως χρειάζεται μία περιορισμένη, αλλά νομίζω αναγκαία αναθεώρηση των συνθήκων. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι σαφές ότι έπρεπε να πετύχουμε μια συνένεση για τον τρόπο εργασίας. Και φτάσαμε σε αυτή τη συνένεση για να εντοπίσουμε εντός των υπαρχουσών συνθήκων πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας Προχωρήσαμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο με συνενετικό τρόπο. Καταρχάς, είπαμε πώς θα βελτιώσουμε τα οριζόντια θέματα και τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Επίσης, μελετήσαμε το πώς θα βελτιώσουμε τις διαθεσμικές σχέσεις τη λειτουργία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελευταίο και σημαντικό, το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Για το πρώτο σημείο. Επικουρικότητα και αναλογικότητα. Η μεγάλη συνένεση στο Συμβούλιο είναι ότι τα εργαλεία για να παρακολουθούμε αυτές τις αρχές τα έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε την συγκεκριμένη λειτουργία. Δηλαδή μια πιο ευέλικτη ερμηνεία της προθεσμίας που δίδουμε στα εθνικά κοινοβούλια για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Περισσότερες ευκαιρίες για τα εθνικά κοινοβούλια για να ασκήσουν εκ των προτέρων ελέγχους για την επικουρικότητα. Η ανάγκη η Κομισιόν να δώσει μεγαλύτερο βάρος στις αιτιολογημένες νομοδοτήσεις, στην περίπτωση ας πούμε της κίτρινης κάρτας. Και η ανάγκη να επιτρέψουμε στα εθνικά κοινοβούλια όχι μόνο να δουλέψουν επί της αρχής της επικουρικότητας, αλλά κάπως να συμπεριλάβουμε και την αρχή της αναλογικότητας στην αξιολόγησή τους. Επίσης, η ανάγκη με βάση το, την άποψη του, του Συμβούλιο να δώσουμε μεγαλύτερο ρόλο στην Κόζακ και προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Κόζακ κατά διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας πιέσαμε ούτω ώστε η Κόζακ να γίνει πιο ενεργή. Αλλά η ατζέντα της μπορεί να εμπλουτιστεί. Διάφορε αντιπροσωπείε επίση κάλεσαν την Κομισιόν μέσω της Προεδρίας να υποβάλει μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίκαιο διοικητικών διαδικασιών. Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε από κάποιους βουλευτές της Επιτροπής ΑΦΚΟ όταν ε, συναντηθήκαμε και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, κάτι τέτοιο θα είναι επωφελές γιατί θα είναι πιο αποτελεσματικά τα πράγματα και θα είναι πιο διαφανής η ευρωπαϊκή διοικητική διαδικασία ή διοικητικές διαδικασίες. Για την, το διαθεσμικό προγραμματισμό Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τον νομοθετικό προγραμματισμό. Είμαστε έτοιμοι για να ενισχύσουμε τη διαθεσμική συνεργασία και να κάνουμε νέες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της διαθεσμικής συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία. Να τροποποιήσουμε δηλαδή τα όσα αποφασίσαμε το 2003, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές οι νομοθετικές εργασίες και να έχουμε και πιο θετικά αποτελέσματα, ούτω ώστε η διαδικασία λήψη των αποφάσεων να είναι πολύ πιο ταχεία. Όσο καλύτερα προγραμματίσουμε τα πράγματα, τόσο πιο ομαλά θα εργαστούμε στα πλαίσια της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας. Επίσης, ως Προεδρία, ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε μια πολιτική δήλωση μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε περισσότερο χρόνο, μας είπε, για το αν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη συμφωνία για τον θεσμικό προγραμματισμό, διαθεσμικό προγραμματισμό. Νομίζω ότι η Λετωνική Προεδρία θα πάρει τη σκητάλη από εμά και θα το, πιέσει, θα το σπρώξει αυτό το σημείο, ούτω ώστε να δούμε αν μπορούμε να υπογράψουμε αυτή την πολιτική δήλωση για το θέμα αυτό. Το άλλο θέμα που αγγίξαμε είναι το θέμα του, της καλύτερης νομοθεσίας. Να συνεχίσουμε δηλαδή το πρόγραμμα REFIT. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να ενισχύσουμε και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της νομοθεσίας με ρήτρε ραντεβού, ούτω ώστε να αποτιμήσουμε το κόστος της μη Ευρώπης, δηλαδή την αδράνεια στο επίπεδο της νομοθεσίας, ε, την έλλειψη νομοθεσίας σε κάποιους τομείς, σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει θέληση στο Συμβούλιο να ενισχύσουμε το ρόλο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ε, προετοιμάζοντας το, τη Σύνοδο και μετά τη Σύνοδο Επίσης θα πρέπει να γίνει μια τακτική συζήτηση για την κατάσταση εφαρμογής των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Κάναμε αυτή την συζήτηση κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας κάθε μήνα. Η Λετωνική Προεδρία και Αντιπροσωπεία, αλλά και άλλες αντιπροσωπείες ε, θεωρούν ότι μη άπαξ του εξαμήνου αρκεί, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε σε ποια φάση βρίσκονται τα συμπεράσματα και κατά πόσο εφαρμόζονται τακτικά, όχι μόνο μία φορά το εξάμεινο. Επίσης θέσαμε το θέμα των διαφόρων μορφωμάτων του Συμβουλίου, των διαφόρων σχηματισμών του Συμβουλίου. Εμεί πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτού του σχηματισμού, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των αντιπροσωπείων δεν πιστεύει κάτι τέτοιο. Πιστεύουν ότι οι σχηματισμοί του Συμβουλίου είναι επαρκεί, είναι ικανοποιητικοί, αλλά υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε κυρίω τη λειτουργία και το ρόλο του Συμβουλίου διαγωνιστικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείναμε επιτυχώς τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα που θα πρέπει να προετοιμάσει καλύτερα και να συντονίσει καλύτερα τις οριζόντιες δραστηριότητες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Εν κατακλείδη, για το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της συνθήκης της Λισαβόνας. Σίγουρα θα πρέπει να διευκολύνουμε τον τρόπο με τον οποίο δρομολογούνται οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών. Η συλλογή των ε, υπογραφών θα πρέπει να γίνεται και ηλεκτρονικά. Να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα εμπόδια που εμποδίζουν τους πολίτες από το να χρησιμοποιήσουν αυτό το 100% δημοκρατικό εργαλείο για τη διαθεσμική συμφωνία που υπογράφεται εκτός του πλαισίου των συνθήκων. Σίγουρα η πρώτη επιλογή ήταν να δουλεύουμε μέσα στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κρατήσουμε τη διαθεσμική συμφωνία που υπογράφεται εκτός των συνθήκων ως εξαίρεση και ως προηγούμενο και όχι ως προηγούμενο ούτως ώστε να ακολουθήσουν και διάφορες άλλες διαθεσμικές συμφωνίες, πολλαπλές ας πούμε, για να αντιμετωπίσουμε άλλα θέματα, τα οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα αντιμετωπίσουμε μέσω των συνθήκων ή μέσω τροποποίηση των συνθήκων. Φερρυπίν, τα διάφορα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση. Εντό των συνθήκων πρέπει να αντιμετωπιστούν και όχι με διαθεσμικέ συμφωνίε. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους και όχι να αποκλείει κάποιους. Θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση της μη συμμετοχής κάποιων κρατών μελών και των πολιτικών επιπτώσεων από την ε, παρακαμψή τους, ας πούμε. Και επίσης, θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητε ολοκλήρωση προσφέρει η συνθήκη των συνθήκων και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό τη. Επίση, υπήρχε κάποιο σκεπτικισμό ε, για το κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιούμε τι διάφορε πασαρέλε, ε, ρήτρε πασαρέλα που έχει το άρθρο 48 48-7. Ο μηχανισμό χρήση αυτών των οδών είναι πάρα πολύ προβληματικό και υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμό για τη χρήση του. Είναι ένα άλλο σημείο το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Αυτά είναι αμυγός θεσμικά θέματα, αμυγός διοικητικά, που συζητήθηκαν στην ομάδα φίλων της Προεδρίας. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, επίσης, Πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την συνθήκη τη Λισαβόνα με συγκεκριμένε πρωτοβουλίε. Παραδείγματο χάρη στην οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση, κάνουμε μια συζήτηση για του αυτόματου σταθεροποιητέ, που είναι ένα εργαλείο αλληλεγγύη, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί μέσα στην ισχύουσα συνθήκη. Είχαμε τη συζήτηση αυτή για τον, το θέμα αυτό τον Ιούλιο και είπαμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για να εφαρμόσουμε πλήρω την αρχή τη αλληλεγγύη στην ισχύουσα συνθήκη και να βελτιώσουμε την οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση. Ένα άλλο θέμα που αναφέραμε στην Προεδρία μας είναι η ανάγκη να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση για την, οικονομική και οικονομική, για την πολιτική και οικονομική ένωση. Και είπαμε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας ότι θα πρέπει να δούμε τα απομεινάρια της σχετικής έκθεσης εφαρμόσαμε μόνο πλήρως την Τραπεζική Ένωση. Καμία άλλη από τις υπόλοιπες ενώσεις, ούτε την πολιτική κτλ. Αλλά μπορούν να γίνουν πάρα πολλά για την δημοσιονομική, το δημοσιονομικό δυναμικό, για την πολιτική ένωση κτλ. Ήταν σημαντικό ότι το η Σύνοδος Κορυφής τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο έδωσε εντολή. Θα συνεργαστούμε με τη Λετωνική Προεδρία για να παρουσιάσουμε τη νέα έκθεση που αναμένεται τον Ιούνιο του 2015 για αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που ήθελα να σας αναφέρω. Και με μεγάλη χαρά τώρα είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ερωτήσεις επ' αυτών των θεμάτων ή επί άλλων θεμάτων. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ευθύ αμέσω δίνω το λόγο στους βουλευτές. Ο κύριος Σέπφλιν. Ευχαριστώ. Ένα θερμό καλώς ορίσατε εκ μέρους του Λαϊκού Κόμματος και εκ μέρους μου κύριε Υπουργέ. Ασφαλώς η Προεδρία σας είναι πολύ δραστήρια και εντυπωσιακό το εύρος των θεμάτων που σας απασχολεί. Και καινοτόμα η προσέγγιση σας. Είμαι βέβαιος ότι και άλλοι συμμερίζονται την άποψή μου όταν λέω ότι αυτά που είπατε, για παράδειγμα, Friends of the Presidency, αλλά επίσης η αύξηση των επενδύσεων και άλλα θέματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θυμάστε όταν μας είδατε πέρσι τον Μάρτιο πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα ακόμη. Είχατε τότε θέσει υπόψη μας έναν αριθμό στόχων μεν, αλλά μάλλον ήταν φιλοδοξίες. Βέβαια τα γεγονότα οδηγούν τους ανθρώπους αλλού. Μια ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι μιλήσατε για τη σημασία της αντιμετώπισης του θέματος της μετανάστευσης. Πού βρίσκεστε τώρα. Δεν είπατε βέβαια και τίποτα για τον κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβαίνουν βέβαια τους τελευταίους 7-8 μήνες πολύ σημαντικά πράγματα όπως στη Μέση Ανατολή, όπως ε, διάφορες ε, ε, εκδηλώσεις τρομοκρατίας. Επίσης Ρωσία, η συμφωνία με τους Αμερικανούς, TTIP. Χαίρομαι που θέσατε και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω η λύση που αναφύεται σιγά σιγά αν δεν έχει λάβει ακόμα τελική μορφή, ε, να διεξάγεται δηλαδή μια τακτική συζήτηση, όπως είπατε εσείς, για κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, για την ποιότητα της ε, δημοκρατίας στο Συμβούλιο έστω μια φορά το χρόνο ή όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο, είναι σωστή λύση. Αντί των εναλλακτικών ε, λύσεων που έχουν προωθηθεί εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέρη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό εξασφαλίζει ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Και βεβαίω είναι δύσκολη, είναι ευαίσθητη η ισορροπία μεταξύ πολιτική και δικαίου. Δεν θα πρέπει να είναι κανεί υπερβολικά βασισμένο ας πούμε, σε νομικίστικα επιχειρήματα, ούτε και υπερβολικά στα πολιτικά. Νομίζω μιλήσατε και για αναθεώρηση των συνθήκων, αλλά βάλατε και ένα ερωτηματικό πίσω. Εδώ έχω ορισμένα ερωτήματα. Θα γίνει σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε το ενδεχόμενο να συγκριθεί μια πανευρωπαϊκή συνέλευση. Μήπως συρθούμε σε μια συνέλευση. Υπάρχουν τόσα θέματα που μας οθούν όντω προς μια κατεύθυνση αναθεώρηση των συνθήκων. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά διαδικαστικά και αλλιώ, αλλά νομίζω ότι σε κάποια χρονική στιγμή θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την αναθεώρηση των συνθήκων. Το ερώτημα είναι, σε τότε εδώ την κοινοβουλευτική θητεία, στην επόμενη, και αυτό που σκέπτομαι είναι εάν πρόκειται να έρθει θα πρέπει να ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση. Και διορτώ με ποιες άραγε είναι η απόφαση σας από αυτού. Τέλος τι γίνεται. Όταν εισήχθη ο θεσμός της Τρόικα έγινε με ε, ιδιαίτερα πανηγυρικό τρόπο. Αλλά τώρα ποιε είναι οι εμπειρίε σα από την Τρόικα. Αξίζει τον κόπο αυτό το όργανο ή αυτός ο θεσμός να υπάρχει και να λειτουργεί. Ο πρόεδρο δεν έχει μικρόφωνο. Ο κύριο υπουργό λαμβάνει το λόγο. Σας ευχαριστώ για τη μετανάστευση. Δεν έφυξα το θέμα αυτό, αλλά για μας Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε στη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών τον Οκτώβρη στο Λουξεμβούργο ήταν θετικό, θετική, θετικό το συμπέρασμα. Βάλαμε μια αρχή σύμφωνα με την οποία τα εξωτερικά σύνορα μια χώρας μέλους είναι κοινά εξωτερικά σύνορα. Ω Ιταλία εμεί επιμένουμε από αυτού εδώ και χρόνια. Για πρώτη φορά όμω υπάρχει ομόφωνη απόφαση των 28 χωρών μελών ότι τα σύνορά μας είναι κοινά σύνορα. Και επειδή είναι κοινά σύνορα, συνεπάγονται συλλογική ευθύνη και κοινέ δράσεις. Βεβαίως, σημαίνει κοινέ επιχειρήσεις. Αυτό, και, αυτό ήταν και αυτό που έδωσε πραγματική υπόσταση νομίζω τα λέει αυτά και το άρθρο 21 της συνθήκης και ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί ως τώρα πριν από αυτήν την επιχείρηση. Το δεύτερο θέμα, για να προχωρήσουμε στη βάση ενός πραγματικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, Απέχουμε βέβαια πολύ ακόμη από αυτό και πρέπει να το θεωρήσουμε προτεραιότητα. Γιατί στην άλλη πτυχή της κοινή πολιτικής μετανάστευσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα πραγματικό κοινό σύστημα ασύλου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο ακόμα πρέπει να γραφτεί μέσα σε αυτήν την ε, κοινοβουλευτική θητεία. Και επίσης το άλλο είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών προέλευσης των μεταναστών. Στις 27 Νοεμβρίου έγινε το 2014 δηλαδή, έγινε σχετική διάσκεψη στη Ρώμη με στόχο να ενισχύσουμε την οικονομική συνεργασία και υποστήριξη και τη συνεργασία στην συνδιαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Γνωρίζετε ότι έχουμε αυτή την συνεργασία για την κινητικότητα. Μέχρι τώρα νομίζω έχουμε μείνει πολύ κάτω από το απαραίτητο και χρειάζεται ενίσχυση. Όμως όλη αυτή η δέσμευση που επιτύχαμε στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας μας για το επιχειρησιακό αυτό πλαίσιο πρέπει πια να εφαρμοστεί. Έχουμε αναπτύξει αυτή την συνεργασία πολιτική μετανάστευσης διαδικασία του Χαρτούμ με το κέρας της Αφρικής και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα. Τώρα, πιο θεσμικά για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας συζητήσαμε την ενδεχόμενη προσφυγή στο άρθρο 31 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορεί μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ το Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Υπάρχει λοιπόν εκεί ανοιχτό ένα παράθυρο για τη χρήση αυτής της πλειοψηφίας, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατεφαρμογή της συνθήκης. Βέβαια συζητήθηκε συζητήθηκαν και άλλοι τρόποι για βελτίωση της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ομάδα επιτρόπων για τις εξωτερικές σχέσεις. Χρειάζεται να βαθύνουμε ακόμη τη συνεργασία μας, χρησιμοποιώντας και τη διαρθρωτική συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουμε διαρκείς δομές συνεργασίες ανάμεσα στις ε, χώρες μέλη που το επιθυμούν και που το δέχονται και να ενισχύσουμε και τον ρόλο της ε, είπα της εκπροσώπου και στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας και αντιμετωπίση των ε, νέων προκλήσεων που έχουν σχέση με την ασφαλειά μας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την ψεύδο διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Ασφαλώς και χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση για τα θέματα ασφάλειας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένα έργο ολοκλήρωσης για τα επόμενα χρόνια, μια πορεία προς την ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι τα θέματα της ασφάλειας. Είχαμε στη δεκαετία του 80 την ενιαία αγορά, στη δεκαετία του 90 το ενιαίο νόμισμα, τώρα εδώ το θέμα που τίθεται είναι η ασφάλεια και επομένω και κράτο δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα πρέπει να είναι αυτό που θα εμφυσίσει ε, ένα πνεύμα και μια έμπνευση στα επόμενα χρόνια. Τώρα πια που δεν είμαι πρόεδρος, σας λέω καθαρά ότι είμαι υπέρ μιας αναθεώρησης των συνθήκων. δηλαδή πλέον δεν δεσμεύομαι από ε, τα δεσμά της Προεδρίας της Ένωσης. Ως μέλος της Ιταλικής Κυβερνήσεως είμαι απόλυτα διατηρημένος να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή σας ειδικά για να εντοπίσουμε τα θέματα που θα πρέπει να επανεξεταστούν, να αναθεωρηθούν στα πλαίσια της αναθεωρήσης αυτής. Νομίζω βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πιο ανοιχτή δημοκρατική μέθοδο που ότως είναι η συνέλευση. Ασφαλώς υπάρχουν ασυνέπειες και φόβοι μεταξύ χωρών μελών στο ίδιο το Συμβούλιο. Έλλειψη συνέπειας εννοώ διότι ορισμένε χώρες μέλη τη Δευτέρα σα λένε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η economic governance, την Τρίτη σας λένε ότι πρέπει να το κάνετε αυτό με την ε, μέθοδο της, ε, του Fiscal Compact, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Την Τετάρτη σας λένε ότι ίσως δεν είναι ρεαλιστικό να μιλεί κανείς για να τι συνθήκες. Κοιτάξτε, τι να σας πω, πώς είναι δυνατόν, μέχρι πού θα φτάσουμε το Σαββατοκύριακο άμα συνεχίσουμε έτσι, γιατί φτάνα, φτάσαμε στην Πέμπτη. Είναι καθαρό πάντως ότι ορισμένα θέματα, ιδίω οικονομικής ε, διακυβέρνησης, αλλά όχι μόνο, και ορισμένα θέματα βιομηχανικής πολιτικής, πολιτικής ενέργειας, εκπαίδευσης παιδείας. Ορισμένα θέματα μπορούν να μπουν στα πλαίσια μιας αναθεώρησης των ε, συνθήκων, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν και κάποιοι φόβοι μέσα στο Συμβούλιο, κάτι που θα συμβάλλει θετικά Εκεί μάλλον θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν σύμφωνα με τι συνθήκε αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει μια αναθεώρηση των συνθήκων, έχοντας βεβαίως συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που δείχνουν τι μπορεί να γίνει με την υπάρχουσα συνθήκη. εφόσον δηλαδή εκμεταλλευτούμε το πλήρε δυναμικό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, συγγνώμη. Αλλά αυτό θα δείξει βέβαια και τα όρια που θέτει η συνθήκη αυτή. Σε ό,τι με αφορά, εγώ θα ήμουν υπέρ μια τέτοια προσέγγιση. Για την τριάδα, το τρίο, μέχρι τώρα η τριάδα ασχολείται μόνο με τον νομοθετικό προγραμματισμό. Κάτι άλλο που μπορούμε ενδεχόμενα να κάνουμε μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθήκων είναι να βελτιώσουμε την συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών της Τριάδας και για ευρύτερα θέματα πολιτικού χαρακτήρα σήμερα περιορίζονται στο νομοθετικό πρόγραμμα. Χρήσιμο μεν, αλλά θα μπορούσε να γίνουν και άλλα πράγματα. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο, δίνει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι η Ιταλική ε, Προεδρία συνέπεσε με μια ιδιαίτερη περίοδο της έναρξης μιας ε, ε, θητείας ε, που σημαδεύτηκε από όλες τις ε, θεσμικές συμφωνίες που συνάφθηκαν. Για μένα απετέλεσε επιτυχία. Είναι σημαντικό το ότι η θεσμική λειτουργία μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του, στα αίτημα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την εκλογή του πρώτου Κομισιόν, σε ό,τι αφορά την πολιτική συμφωνία που αντικατοπτρίζε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ε, της ακροάσης καινούριας επιτροπής κλπ. Πιστεύω ότι η μεγάλη πολιτική επιτυχία αυτής της περίοδου ήταν το ότι η Ευρώπη μετά τις τελευταίες ευρωεκλογέ ξεκίνησε με το δεξί ας πούμε. Επίσης ε, είχατε και συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Δυστυχώς όμως είναι θέματα που αυτή τη στιγμή δεν συζητώνται πάρα πολύ στην Ευρώπη. Όμως τους τελευταίους τρεις μήνες ιδιαίτερως, όχι μόνο με το σχέδιο Juncker, αλλά και με τις ε, πολιτικές συμφωνίες για την ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας, ε, με τις κινήσεις του κυρίου Ντράγκη στην ΕΚΤΑ. Όλα αυτά φαίνεται να σηματοδοτούν μια αλλαγή πορείας της ε, Ευρώπης που επιθυμούμε. Θέλω όμως να θέσω και ένα σημαντικό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Το πιο αρνητικό συμβάν κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας ήταν η είδηση ότι τα ευρωπαϊκά κράτη σε φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα είμαστε ε, μια καταστροφή. Υπάρχει μια έλλειψη ε, φορολογικής και δημοσιών, φορολογικής βασικά ε, αλληλεγγύης και δεν μιλούμε μόνο για τα LuxLeaks που ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Ε, υπάρχει ένα αίτημα φορολογικής δικαιοσύνης αφενός, ε, αυτό είναι σίγουρο, αλλά υπερβαίνει αυτό το ζήτημα το πρόβλημα. Πρόκειται για την εναρμόνιση των φορολογικών μας συστημάτων, πρόκειται για το συντονισμό στην παροχή φορολογικών πληροφοριών, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό φορολογικό ε, σύστημα. Ε, η ομάδα των σοσιαλιστών δεν θέλησε ε, να συμμετάσχει σε πολιτικές κινήσεις που θα αποσταθεροποιούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να συνεργαστούν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, ο κύριος Γιούγκερ ανέλαβε συγκεκριμένε δεσμεύσει ε, ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο. Αλλά και το Συμβούλιο ε, πρέπει να κάνει κάτι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δουλειά του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, την ε, επόμενη Προεδρία. Πώς ε, εργάζεται το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ώστε να δώσει μια ταχεία απάντηση στα αιτήματα των πολιτών να λαμβάνει χώρα φορολογική, φορολογικό συντονισμός και μια φορολογική και να υλοποιηθεί προοδευτική, συγγνώμη, φορολογική προοδευτικότητα στην Ευρώπη. Ε, την ανησυχία σας Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας δουλέψαμε πολύ για αυτό το θέμα και πετύχαμε σημαντικά θε... Ε, αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών ανάμεσα στις ε, κυβερνήσεις. Πείσαμε ιδιαίτερως δύο κράτη-μέλη που ιστορικά διαφωνούσαν με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών να ε, ενταχθούν σε αυτό το σύστημα από το 2017 και μετά. Θα είναι ένα πραγματικά καλό εργαλείο που μας έλειπε προκειμένου να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Η Νέα Επιτροπή Juncker ε, θέλει να προχωρήσει το θέμα της ε, φορολόγησης των επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Ο φορολογικός ανταγωνισμός Ε, δεν ήταν ποτέ ε, οικονομικά δεκτός, τώρα πια δεν είναι ούτε κοινωνικά αποδεκτός. Ε, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ε, παραβιαστεί και η αρχή της εμπιστοσύνης στην συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση ό,τι αφορά την αμοιβή εμπιστοσύνη. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ε, των μέτρων που έχουν δημιουργήσει αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης στην οποία θα πρέπει να, στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε. Επίσης υπάρχει και το εμπόδιο της ομοφωνίας. Ακόμα και όταν ε, επιλέγουμε τον δρόμο της ενισχυμένης συνεργασίας πάλι δεν έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Το, στο θέμα του φόρου των ε, συναλλαγών ε, επιλέξαμε αυτό το δρόμο ε, της ενισχυμένης αλλά και πάλι δεν έχουμε ακόμα αυτά αποτελέσματα. Απ' την άλλη μεριά οι πολιτικές δεσμεύσεις της Κομισιόν είναι πολύ σημαντικές αντικατοπτρίζονται στο νομοθετικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς και θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Κύριε. Μπρέσο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. όχι τόσο ως Ιταλίδα θα μιλήσω, αλλά ως υπέρ, ως ε, θειασότρια του φεντεραλισμού. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν ως φεντεραλίστε για όλα όσα μας είπατε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση που κάνατε για πολλά σημεία και στα οποία μπορούμε να επανέλθουμε σε ό,τι αφορά κυρίως το δυναμικό της Λισαβόνας. Στο δεύτερο κομμάτι της θητείας μας μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για την πολιτική ενότητα της Ευρώπης. Νομίζω ότι ε, με τα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο είναι όριμη αυτή η συζήτηση. Ε, και συνδέεται και με το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Υπ' αυτή την έννοια το δυναμικό της Λισαβόνας είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που ισχύζονται συχνά οι σχολιαστές. Και αυτό το έδειξε. Η δράση που είχαμε για το θέμα της εκλογής του Πρόεδρου της Κομισιόν που οδήγησε σε αυτό το σχέδιο για τις επενδύσεις που άνοιξε ένα δυναμικό έμεσης λήψης χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς... Σύναψης χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η πολιτική κατεύθυνση που παίρνει το Συμβούλιο υπό την έμπνευση και καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και είναι σημαντικός και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις δυνατότητε που του δίνουν οι συνθήκες και αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ακόμα που θα μπορούσα να πω, αλλά ένα είναι σημαντικό, ιδιαίτερο σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα που συνδέεται με την Λισαβόνα, χρήση της Λισαβόνας και μια νέα ενδεχόμενη συνθήκη. Το θέμα της άμυνας και ασφάλειας Ευρώπης. Φαντάζεστε ότι σήμερα το θέμα αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες και μπορεί να ξαναδώσει στην Ευρώπη αυτή την νομιμότητα που κάποιοι θέλουν να τις αφαιρέσουν. Και αυτό το θέμα μπορεί να, αυτός ο τομέας μπορεί να ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στη συνθήκη. Θα ήθελα εδώ να μου κάνετε μια αξιολόγηση. Πιστεύω μια, ότι μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αναλυθεί από κοινού ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αν στα πλαίσια των συνθήκων μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη κοινή ασφάλειας και άμυνας. Και εν πάση συνεχεία να δούμε και ποια θέματα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια νέα συνθήκη. Ας ε, πούμε ποια είναι η δυναμική Τη Λισαβόνας, η σημερινή δυναμική τη Λισαβόνας, ποια θέματα μπορούν να ενταχθούν εκεί και τι μπορεί να μπει σε μια νέα συνθήκη. Κοιτάξτε, πριν από εσά ε, ήρθαν κάποιοι νέοι εδώ και μίλησαν. Δεν ήσασταν ακόμα εδώ. Οι νέοι μας κάλεσαν να βρούμε το θάρρο για να προτείνουμε ένα βασικό νόμο. Το θέμα της νέας συνθήκης δεν να μην συνδέεται μόνο με συγκεκριμένα θέματα, αλλά να επανέλθει στην αρχική ιδέα της συνταγματικής συνθήκης και να έχει και κάποια συμβολικά στοιχεία κλειδιά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Eh, Μιλάμε για ένα θεμελιώδη νόμο ή για μια συνταγματική συνθήκη με λίγα άρθρα για κοινούς στόχους και συνεχεία να έχουμε παράλληλα πιο λεπτομερή έγγραφα που θα αφορούν τους ενδιαφερόμενους και τους ειδικού. Να δοθεί μια εντολή όχι μόνο για σημαντικά επιμέρους σημεία για τη λειτουργία της Ένωσης, αλλά να δώσουμε κάποια κοινά στοιχεία για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, το ευρωπαϊκό σχέδιο. Να μην μιλήσω για σύνταγμα γιατί είναι φοβιστερή λέξη, αλλά κάτι βασικό. Κάτι που να είναι κοινή κληρονομιά των Ευρωπαίων πολιτών και να το καταλαβαίνουν όλοι μονοσήμαντα. Επειδή θα είναι τόσο απλό και τόσο θεμελιώδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μπρέσκο για το θέμα της αναθεώρησης των συνθήκων. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα ταμπού. Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί και αυτό το θέμα, μια ενδεχόμενη αναθεώρηση. Οι πολιτικοί, οι διπλωμάτες φρικάρουν κάθε φορά που μιλάμε για αναθεώρηση των συνθήκων. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε ανάλογα με τους πολιτικούς μας στόχους. Αν είναι τέτοιοι πολιτικοί μας στόχοι και αν έχουμε την πολιτική ε, θέληση ε, να πάμε σε ε, τομεί, σε παιδεία κτλ. που απαιτούν αναθεώρηση των συνθήκων, γιατί όχι. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου πρέπει να το ξαναδείτε αυτό το θέμα. Ε, σε ό,τι αφορά τη, θεσμική και πολιτική βούληση, ε, νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχά υπάρχει το Fiscal Compact, το δημοσιονομικό ε, σύμφωνο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Και θα δούμε τι αξιολόγηση θα προκύψει. Πρώτα θα πρέπει να αξιολογηθεί και μετά θα πρέπει ενδεχομένω να ενταχθεί σε συνθήκε. Εάν δεν κάνω λάθος, ε, θα πρέπει να ενταχθεί σε μια συνθήκη μέχρι το τέλος του 2017 ή το 2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενσωματώσουμε τις συνθήκες, θα τις ανοποιήσουμε ή θα τις αναθεωρήσουμε. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την λεγόμενη διακυβέρνηση της Νομισματικής Ένωσης. Δεν είναι ούτε δουλειά μου ούτε μπορώ να κάνω προφητείες. Πώς θα πάνε ας πούμε, οι Βρετανικές εκλογές, δεν έχω ιδέα. Αλλά νομίζω ότι η σημερινή η Βρετανική κυβέρνηση είπε ξεκάθαρα ποια θα είναι η διαδρομή. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό από τις εκλογές, τότε θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πρέπει να αρνηθούμε να ανοίξουμε τα αυτιά μας για την ε, Βρετανική συζήτηση, στη Βρετανική συζήτηση, θα πρέπει να τη φοβόμαστε, λάθος θα ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Πρέπει, νομίζω, να συζητήσουμε ε, την αναθεώρηση των συνθηκών, γιατί η πολιτική μας εξωθεί να το κάνουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε, θα αποκόψουμε την πραγματικότητα και την πολιτική συζήτηση από τον ιονή κόσμο, τον φαντασιακό κόσμο, τον ευρωκομμουνιστή ε, τον ευρωκοινοτικό κόσμο, ας πούμε, που είναι φαντασιακός. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τις ασυνέπειες των ε, κρατών μελών που λένε Δευτέρα, Α, Τρίτη, Β και ούτω καθεξής. Δεν το καταλαβαίνω. Ε, επίσης, και από τις εθνικές αντιπροσωπείες ακούω διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνω την ανησυχία ε, κάποιων άλλων κρατών μελών που έγιναν δύσκολα δημοψηφίσματα ή θα γίνουν. Τι θέλουμε, να αποκοπούμε από την πραγματικότητα, να μην λάβουμε υπόψη αυτές τις δυσκολίες. Δεν είναι δυσκολίες όμως που πρέπει να μας αποτρέψουν από την ανάγκη της συζήτηση. και ενδεχομένως την αναθεώρηση των συνθήκων για να υλοποιήσουμε του στόχου μας. Τους μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τι επενδύσει επενδύσεις και την ευελιξία δεν θα επανέλθω, συμφωνώ. Για το θέμα μια ευρώπη. ε, μιας ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Πρέπει να δούμε πότε θα δρομολογήσουμε αυτή την προσπάθεια με ισορροπημένο τρόπο. Ε, ασφάλεια και δικαιώματα, έτσι, και ποια είναι η ισορροπία τους. Οι διαρθρωμένες συνεργασίες ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, με, με μια νέα αντίληψη για την ασφάλεια, που θα συμπεριλαμβάνει και τις εσωτερικές υποθέσεις και τις εξωτερικές υποθέσεις και τις ε, ε, δημόσιες ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ούτε ώστε να τη δώσουμε έτσι μια απτή έννοια για τους πολίτες. Και στο παρελθόν, ε, όταν οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζαν απειλές, βρήκαν το θάρρος για να προχωρήσουν προς αυτή την Ένωση. Είναι κάτι που αναμένεται. Όχι κάτι που θα κάνει η Ευρώπη μέσω των συνθήκων. Αυτό που αναμένεται πάνω απ' όλα είναι, μεγαλύτερη ασφάλεια. Μια εθνική προσέγγιση ασφάλειας και μόνο είναι ανεπαρκής. Αν συνεχίσουμε προς αυτή την ατραπό και το μόνο που μας ενδιαφέρει να προσπιζόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, δεν θα έχουμε ούτε εθνική κυριαρχία, ούτε ασφάλεια θα έχουμε. Ούτε ασφάλεια για τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση. Είναι μια ευκαιρία. Και το λέω εντό αγωγικών βέβαια, έτσι. Εγώ εξεπλάγην από το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά η Ήπειρός μα η Ευρώπη που γεννήθηκε από τα ερήπια του Auschwitz έγινε στο Παρίσι αυτή η απόπειρα στο Σαλί Εμπτό. έγιναν οι επιθέσει αντίον των Εβραίων. Αισθάνονται ανασφαλεί οι Εβραίοι που σκέφτονται, τόσο που σκέφτονται να εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Υπάρχει, μια, ε, υπάρχει τρομοκρατία, υπάρχει μεγάλη Ισλαμοφοβία. Απέναντι όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση. Δεν αρκεί η εθνική απάντηση. Ούτως ή άλλως η απειλή είναι πολύ μεγάλη για τις πόλεις μας, τις ευρωπαϊκές πόλεις. Και αυτό σημαίνει και διαφθομένη συνεργασία και πολλά πράγματα. Άλλα πράγματα. Στο εσωτερικό λοιπόν της ασφάλειας πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο στην ε, ΚΕΠΑ και στην ε, ΕΠΑ περισσότερο την ε, πλειοψηφική ψήφο. Να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο δηλαδή τη συνένεση και την αναζήτηση πλειοψηφίας και να παρακάμψουμε την ομοφωνία. Και αυτό πρέπει να το δούμε και πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις διατάξεις που έχουμε για τις με τη μετανάστευση, πώς θα προωθήσουμε παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα, αυτό που είπατε για το θεμελιώδη νόμο, ένα πανευρωπαϊκό νόμο, το εύχομαι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα όμως και οι ισορροπίες στο Συμβούλιο, δύσκολο μου φαίνεται να φτάσουμε σε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν, σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των κυβερνήσεων για ένα νέο θεμελιώδη νόμο. Τώρα, αν με ρωτάτε αν έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός ή ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με τη Λισαβόνα, κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Έχουμε το, τους νέους εθνικισμούς, έχουμε την Ισλαμοφοβία, τον νέο ρατσισμό κτλ. Ποια είναι η απάντησή μας στην Ευρώπη. Είμαστε λιγάκι λιγότερο ε, φεντεραλιστές, λιγότερο υπέρ της ε, ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Υπό την πίεση της ε, κοινή γνώμης νομίζω ότι αν υποχωρήσουμε αρχίζουμε να συγκεντρώνουμε τα συστατικά για έναν ακόμα πάταγο ας πούμε, για μια ακόμα ευρωπαϊκή καταστροφή. Μία ακόμα ερώτηση από τον Πέντρο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ Σάντρο που είσαι ξανά μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για το πρέμα συνεργασίας που έδειξες με την Επιτροπή μας και συνολικά ευχαριστώ την Ιταλική Προεδρία για τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ιταλική Προεδρία σίγουρα έκανε τη διαφορά. Στήριξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την όθησε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλά σημαντικά βήματα έγιναν. Το επενδυτικό πρόγραμμα, η ανακοίνωση για την ευελιξία. Παρόλο ότι είναι πράγματα που αποτελούν ένα πρώτο βήμα, παρόλο ότι θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Είναι αποτέλεσμα όλα αυτά πολιτικής πίεσης και πιστεύω ότι η Ιταλική Προεδρία έπαιξε σοβαρότατο ρόλο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και την Ιταλική Προεδρία και τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και ό,τι αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναθεώρηση της θεσμικής λειτουργίας και της εργασίας της ομάδας των φίλων της Προεδρίας, καθώς επίσης και τη συζήτηση για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης. Ε, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά πρέπει να δούμε το μέλλον. Η Ιταλία δεν έχει ακόμα την... Δεν έχει πια την Προεδρία. Οπότε απελευθερώθηκε ε, και εσείς ο ίδιος απελευθερωθήκατε από την Προεδρία όπως είπατε. Οπότε μας αναφέρατε τις δικές σας πολιτικές, προσωπικές πολιτικές απόψεις για την αθεώρηση της συνθήκης. Είπατε, σχολιάσατε μάλλον και τις προτάσεις Κομισιόν για την ε, δημοσιονομική ευελιξία και, και το επενδυτικό πρόγραμμα και ταμείο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα ήθελα να ακούσω ε, μια πιο λεπτομερή άποψη από εσάς για αυτά. Ε, βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα, θα γίνεται συζήτηση. Για παράδειγμα, η επενδυτική ρήτρα φαίνεται ότι θα είναι πολύ κοντά να ενταχθεί στο σκέλος, το διορθωτικό σκέλος. Είναι σωστό αυτό. Είναι σωστό να πούμε ότι ε, οι συνεισφορές ενός μέλους που είναι στο διορθωτικό σκέλος στο επενδυτικό ταμείο δεν προσμετρώνται στο έλλειμμά του. Ε, αν όμως είναι στο άλλο το προληπτικό σκέλος προσμετρώνται. Έχει νόημα να πούμε κάτι τέτοιο ήσασταν σαφείς για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αθεώρηση της συνθήκης. Θα ήθελα όμως να μου δώσετε μερικές εξηγήσεις σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα βελτίωση της δημοσιονομικής ευελιξίας που έχει προτείνει η Κομισιόν. Παύλο Ράντζελ και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Θέλω να θίξω ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία και η στάση μας εναντί της Ρωσίας. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προετοιμάζει μια χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον της ε, Ρωσίας. Είδαμε τις τελευταίες μέρες ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιες εξελίξεις, κάποιες κινήσεις. Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον. Είναι σημαντικό γιατί και η, γιατί η Ιταλία θεωρείται πιο ρωσόφιλη από ό,τι άλλες Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ε, Όπως ε, και με την ε, εξετάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτήσεις για όλα τα θέματα. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα. Ε, κάνουμε προσεκτικά βήματα. Αυτά τα βήματα που αναφέρατε είναι προσεκτικά βήματα και για τους συντρικούς μπροστά. Προς τα μπρος. Και είναι βήματα διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί σε ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα. Και σε αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να συμπεριλάβει και την ρήτρα σε ό,τι αφορά τις εθνικές συνεισφορές στο κεφάλαιο του ε, επενδυτικού ταμείου. Η σημασία αυτής της ρήτρα ξεπερνάει τα θέματα λειτουργίας του ε, επενδυτικού σχεδίου. Η αρχή είναι ότι δεν είναι κακές όλες οι δημόσιες δαπάνες. Υπάρχουν και καλές δημόσιες δαπάνες και δημόσιες δαπάνες οι οποίες προορίζονται, συνεισφέρουν στην επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου και που ε, γίνονται από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καλές και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να θεωρούνται ουδέτερες σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας, το σύμφωνο ε, ανάπτυξης. Αυτό είναι ε, επανάσταση σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει για μια επενδυτική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ δε περισσότερο να μιλήσουμε για την ουδετερότητα των εθνικών συνεισφορών. Είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, είναι ανοιχτά. Και δεν μιλώ αυστηρά από την Ιταλική πλευρά, μιλώ λαμβάντας υπόψη όλη την Ευρώπη. ο περιορισμός αυτής της ρήτρα ε, μόνο στο διορθωτικό σκέλος είναι μια πολύ προσεκτική ε, προσέγγιση. Ίσως θα μπορούσαμε να διευρύνουμε την εφαρμογή και στα δύο σκέλη. Δεύτερον, τι θα γίνει με την διακυβέρνηση, ποιος θα είναι ο ρόλος των κρατών μελών στην λήψη των αποφάσεων. Ποιο θα είναι ο ρόλος των εθνικών τραπεζών και των άλλων εθνικών φορέων που θα συμμετάσχουν. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι και αυτό ανοιχτό θέμα. Το βασικό συστατικό για την επιτυχία του επενδυτικού αυτού σχεδίου θα είναι ε, η υλοποίηση μόνο των πιο ελκυστικών ε, σχεδίων. Γιατί αυτά τα ελκυστικά σχέδια κινητοποιούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι σε ορισμένου τομεί που ε, δεν είναι οι πιο αγαπητοί των ιδιωτικών επενδυτών, των ιδιωτών επενδυτών, να μπουν χρήματα. Για παράδειγμα, εκπαίδευση, κοινωνία τη Γνώση κλπ. Επίση, θα πρέπει να επικρατήσει και κάποια ε, γεωγραφική ισορροπία. Αυτή δεν μπορεί να μπει με καθαρούς όρους στο χαρτί, αλλά σίγουρα ένα από τα κίνητρα για να επενδύσει κάποιον, κάποιος θα είναι ε, να υιοθετηθούν και να ελοπιθούν προγράμματα σε συγκεκριμένους κλάδους και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενδεχομένως διασυνοριακές περιοχές. Το σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία. Στο τελευταίο Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων επιμείναμε ότι πρέπει να ε, γίνει εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ με απτά βήματα και ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την ε, έναρξη της μεταρρυθμιστικής εσωτερικής εθνικής διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία. Και τα δύο αυτά παράλληλα. Μετά οι κυρώσεις. Οι δεν αποτελούν αυτό σκοπό, είναι ναι, ένα εργαλείο και ως εργαλείο θα πρέπει να συνοδεύουν σε κάθε στιγμή ε, την, το στάδιο της εφαρμογής κάθε φορά της ε, συμφωνίας του Μίνσκ και το στάδιο υλοποίησης των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων της Ουκρανίας. Αυξομοιούμενες. Ευχαριστώ δεν θυμούμε άλλον υπουργό άλλη προεδρία να είναι προετοιμασμένο να απαντήσει σε τόσο ευρύ φάσμα ερωτήσεων. Όμω σα ζητήσαμε να έρθετε γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είστε μόνο υπουργό, είστε και εμπειρογνώμων. Και γι' αυτό χαιρόμαστε για την συνεργασία μαζί σα. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να έχετε πάντα στα χέρια σα τα σημαντικά θέματα. Πολλά πράγματα μένουν να γίνουν ακόμη στην Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε και πάλι.